Okay, colleagues. Συνάδελφοι. Can I bring the meeting to order the next... Ας ξεκινήσουμε. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν υπάρχουν. Οπότε περνάμε γρήγορα από αυτό. Πάμε στην ψηφοφορία. Πρόταση κανονισμού που τροποποιούν τον κανονισμό 443 καθορίζονται οι τρόποι να, να πετύχουμε τους στόχους του 2020 για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακου στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Πρώτα τα αυτοκίνητα και μετά τα μεγαλύτερα οχήματα. Να ελέγξουμε τα μηχανήματα, οι πληροφορίες, το ηλεκτρονικό μηχάνημα. Βάλτε την κάρτα μέσα παρακαλώ. Βάλτε την κάρτα. Λοιπόν όλοι, βάλτε τις κάρτες. And can you press a button? Πατήστε ένα κουμπί, οποιοδήποτε κουμπί, δοκιμή είναι. Πατήστε ένα κουμπί. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Τελειώσαμε με αυτό. Όλοι είναι εντός των ποσοστώσεων, οπότε ξεκινάμε. Οι μεγάλες ομάδες, κύριε Λίχτεμπεργκ, προσπαθούν να έχουν κάποιον παραπάνω. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές, ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52, 53, 54, 34, 35, 36, μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 και 70 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 και 4 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πάμε στην 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 και 5 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ υπέρ 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 38 ξεκινάει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι το ΕΛΚ έχει έναν παραπάνω ψηφίσατε όλοι πέρας 14 ψήφοι υπέρ, 28 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εκδυνάται. Τελική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. ΕΛΚ ξανά έχει μια ψήφο παραπάνω. Τέλος. 37 υπέρ, 5 ψήφια εναντίον, καμία εποχή, οπότε εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περιμένουμε λιγάκι να βάλω γάλα. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 34 και 21 μαζί υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Σας παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία για την 34 και 21. Το S&D έχει μια ψήφο παραπάνω. Καλώς, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ, 17 εναντίον, εγκρίνεται. 37 και 39 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 38 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει ένα ψήφο παραπάνω. Πέρας. Απορρίπτεται. 21-21. Πάλι καλά που παρακολουθώ τις δύο μεγάλες ομάδες. 36 υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος για το 36. Ξεκινάει 20 έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 21-21. 40 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 40 ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 24-18 Επειδή κρίθηκε η τροπολογία 40, έχουν προφορική τροπολογία του εισηγητού και διαβάζω αύξηση των, του στόχου ειδικών εκπομπών που απορρέει από την εφαρμογή των πολυπεσιαστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα έχει ανώτατο όριο στα 3,5 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος ανά χιλιόμετρο, ανά έτος, ανακατασκευαστή. Ελπίζω κάποιος άλλος εκτός από μένα κάτι να πιάσει από όλα αυτά που είπα. Ε, κύριε Σιγητά, θέλετε να εξηγήσετε τα συντομία και μετά θα ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσεις ο Εισηγητή. Ευχαριστώ. Η τροπολογία που μόλι συγκρίναμε αναφέρεται στα πιστοτικά υπερμόρια. Για να είμαστε λοιπόν συνεπεί με αυτά που ψηφίσαμε στην προηγούμενη γραμμοδότηση, που έχουμε τα πιστοτικά υπερμόρια, αλλά εκεί περιορίζουμε την, ε, την επιδότηση στο 2,5 γραμμάρια, θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε και την συγκεκριμένη γραμμοδότηση σε ό,τι αφορά τα υπερμόρια. Να περιορίσουμε δηλαδή αυτή την επιβράβευση στο όριο των 2,5 γραμμαρίων για να έχουμε ίδια προσέγγιση και στις δύο γραμμοδοτήσεις, δηλαδή και στα ελαφρά φορτηγά και στα επιβατικά. Καλώς, άρα πρόκειται περί συμπληρώσεως. Και πού πάει? Άρα είναι προσθήκη στην τροπολογία 40 που μόλις εγκρίνατε, εντάξει. Υπέρ. Ε, μάλλον, υπάρχουν αντιρρήσεις πρώτα απ' όλα. Ματιό. Ήθελα μόνο να πω πως ε, πρέπει να το ψηφίσουμε, αλλά εγώ προτείνω στο ΕΛΚ να μην το υπερψηφίσει. Ναι, ναι, κατανοητό. Αλλά δεν έχεις αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία. Καλώς. Αυτή η προφορική τροπολογία ως προσθήκη στην τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές θα γίνει έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος. Το ΕΛΚΑ έχει έναν παραπάνω που ψηφίζει. Ψηφίσατε όλοι, πέρας 16 υπέρ, 25 ψήφια εναντίον. Απορρίπτεται. Και πάμε στην τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 42 νομίζω ότι απορρίπτεται άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 13 υπέρ, 27 ψήφοι εναντίον, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 και 52 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Ξεκινάει ο έλεγχος για τη 16. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 33 ναι εγκρίθηκε. Μετά στην επόμενη 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 27 ξεκινάει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε Απορρίπτεται. 15-25. Τελική ψηφοφορία που ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε ένα ΕΛΚ περισσότερο και ένα σωσιαστή παραπάνω. Τώρα είμαστε εντάξει, πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται 36 με 5. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και για τις δύο εκθέσεις. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Η κυρία Τσικάου κανονικά θα μας ενημερώσει, αλλά την περιμένουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τη Σίλβια για τις ταχυγράφους. Τι γίνεται στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ε, Τετάρτη που μας ε, πέρασε 20 Μαρτίου συζητούσαμε στον τριμερή διάλογο τον ψηφιακό τάχογράφο με την Προεδρία προχωρήσαμε πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο ξεκαθάρισε αρκετά βεβαίως υπό την προϋπόθεση πως θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατάφεραν να βελτιώσουν το κείμενο της ε, Κομισιόν Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τη Γραμματεία για την πάρα πολύ μεγάλη στήριξη που έχουμε συνεχώς και βεβαίως ε, τον ε, σκιώδη και τους σκιώδη και τους συνεργάτες της ομάδας μου. Λοιπόν, βελτιώσαμε την ε, πρόταση, πολλές προτάσεις κομισιών και καταφέραμε παραδείγματο χάρη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στα θέματα των νέων λειτουργιών των ψηφιακών ταχογράφων να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο, δηλαδή νέες λειτουργίες, ε, προειδοποιήσεις, ε, το τι γίνεται με τα καταγεγραμμένα δεδομένα, όλα αυτά μπήκαν σε ένα νέο άρθρο. που έχουμε την τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες πλέον αντικατοπτρίζονται σε αυτό το άρθρο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, νέα μέτρα για να υπάρξει ένας ανοιχτός ανταγωνισμός όσον αφορά την εμπορία αυτών των ταχογράφων και βεβαίως βελτιώθηκε, βελτιώθηκαν και αυτά τα οποία φορούσαν τα των ελέγχων και των φορέων που θα κάνουν τσε, ε, τους ελέγχους αυτούς και υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, που αφορούν ε, την ε, κοινή ερμηνεία της ε, κοινωνικής ε, νομοθεσίας. Κατόπιν έχουμε την το τι γίνεται με τα τελείως νέα φορτηγά και αυτά τα οποία θα εξοπλιστούν εκ των υστέρων με τέτοιον εξοπλισμό. Το Κοινοβούλιο οπωσδήποτε προσπάθησε πάρα πολύ για να επιτύχουμε κάποιες ε, καλύτερες διατάξεις στο ζήτημα της ε, κοινωνικής ε, νομοθεσίας και ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί η Προεδρία ήδη από την αρχή ήταν πάρα πολύ αρνητική όσον αφορά τα κοινωνικά. Και πήγαινε πιο πέρα από την Κομισιόν και η Κομισιόν ήταν εναντίον των ε, ε, θέσεων του Κοινοβουλίου αλλά καταφέραμε να αποσπάσουμε μία δήλωση για μία αναθεώρηση του κανονισμού του 2006 και σε σχέση με την δυσκολία των διαπραγματεύσεων εγώ ως εισηγήτρια φρόντισα να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και η δυνατότητα κάποιων εξαιρέσεων στην χρήση των ταχογράφων αυτών σε μικρά φορτηγά κάτω από 7,5 τόνους και όταν μιλάμε για διαδρομές οι οποίες δεν είναι εμπορικές με την συνήθεια έννοια και επίσης τα 107 χιλιόμετρα γύρω από την έδρα της εταιρεία αναφέρθηκαν και αυτή είναι η μοναδική δυνατότητα που υπάρχει να συμπεριληφθούν οι μη επαγγελματίες οδηγοί, αυτοί οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα σε μία εξαίρεση, κάτι το οποίο ζητούσε οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο, σημαντικό, είναι πως ε, θα έπρεπε οι αρχές που κάνουν τον έλεγχο να μπορούν να ελέγχουν ε, του μακρόθεν τα οχήματα αυτά, τον ταχογράφο αυτων Η Προεδρία είπε πως εδώ πέρα υπάρχουν σοβαρές αντιστάσεις για το ζήτημα αυτό, γιατί μας είπαν πως θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Και έχουμε οικονομική κρίση κτλ. Αλλά εγώ τους είπα, μα οικονομική κρίση δεν έχουν μόνο τα κράτη-μέλη, έχουν και οι μεταφορικές επιχειρήσεις. Οπότε είναι δύσκολο να απαιτήσουμε από τις επιχειρήσεις να βάλουν καινούριου ψηφιακούς ταχογράφους και τα κράτη-μέλη να μην κάνουν καμία επένδυση ε, και να μην κάνουν τουλάχιστον ε, αυτή την ε, βασική επένδυση. Τέλος, ήταν και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση στο θέμα των πράξεων κατεξιοδότηση. Ήδη ήταν σαφές ε, ευθύς εξ αρχής πως ε, Δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο για τις τεχνικές λεπτομέρειες. θα, έπρεπε βεβαίω κάτι τέτοιο, να, οτιδήποτε προβλεφτεί να είναι νόμιμο και να διαφυλάσει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Οπότε γίνεται η προσπάθεια έτσι ώστε να μπουν στο δυνατόν περισσότερες διατάξεις ε, στον βασικό κανονισμό που θα είναι στην συναπόφαση. Αναμένοντας λοιπόν τον επόμενο γύρο τριμερούς διαλόγους στις 6 Απριλίου θα συζητηθούν δύο ακόμα θέματα. Δηλαδή το ότι δεν θα σβήνει αυτόματος στοχογράφος όταν σβήνει ο κινητήρας και δεύτερον το ότι για οδηγούς που δεν έχουν την έδρα τους ε, σε μια χώρα θα υπάρχει μια προσωρινή, ε, ένα προσωρινό τέτοιο μηχάνημα που θα λειτουργεί για 58 ημέρες. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν εάν το Συμβούλιο δεχτεί τα άλλα δύο βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου και υπάρξει τουλάχιστον ένας ελάχιστος εξοπλισμός με τα μηχανήματα αυτά τα οποία ζητήσαμε και να μην εξαιρούνται οι επαγγελματίες οδηγοί όταν ε, είναι στο... στην ακτίνα των 100 ε, χιλιόμετρων από την έδρα της επιχείρησης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τους κοιοδησηγητές και τους ε, Ωραία, να σα υπενθυμίσω ότι αν υπάρχουν απορίε ή ερωτήσει, ευχαρίστω να τι απαντήσουμε, αλλά δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση, γιατί έχουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή είναι ε, σημαντική. Αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις απορίε, πολύ ευχαρίστω. Αν ε, διαπιστώσω ότι κάποιο αρχίσει και κάνει συζήτηση και παρατηρήσει, θα κόβω το μικρόφωνο. Λίχτεμπεργκερ και μετά ο κύριο Πίρκερ. Ja, und genau das möchte ich auch tun. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια η οποία πραγματικά παλεύει ως Λένα, σαν Λένα για την θέση του Κοινοβουλίου και πραγματικά η στάση του Συμβουλίου εδώ πέρα είναι σκανδαλώδη γιατί θέλει δύο πράγματα. Είτε ένα κανονισμό που θα έχει τόσα παραθυράκια που δεν θα σημαίνει τίποτα είτε να μην οδηγηθούμε πουθενά. Δηλαδή σε μια ρύθμιση η οποία νομοθετικά δεν θα στέκει. Είναι σκανδαλώδες αυτό το οποίο κάνει το Συμβούλιο. Είναι χαστούκι στο πρόσωπο οποιοδήποτε ξέρει λίγο αυτά τα πράγματα και πρέπει να σας πω ειλικρινά πως έτσι πρέπει να τα πούμε ομά, γιατί εδώ πέρα ε, το Συμβούλιο μας εκβιάζει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Κύριε Πέρκερ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις. Γιατί δεν άκουσα ακριβώς πώς έχουν οι ε, αυτό με τις ε, μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και τα λοιπά, ε, σωστό και σας ευχαριστώ. Εκεί πέρα αντιλήφθηκα πως ε, πράγματι θα πάει στην κατεύθυνση αυτή που αναφέρθηκε με τα 100 χιλιόμετρο και η δεύτερη εξαίρεση αφορά το άρθρο 13 όπου λάβαμε μία απόφαση ως Επιτροπή να εξαιρέσουμε και τις ε, παραδόσεις οικοδομικών υλικών στα εργοτάξια. Από αυτό δεν άκουσα τίποτα από την εισηγήτρια, θα ήθελα να ακούσω κάτι. Και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή αναφέραμε και τους 3,5 ε, τόνους αντί για τους 2,8. Πώς έχει εκεί η διαπραγμάτευση. Μάλιστα, πριν απαντήσει η εισηγήτρια, δεν θέλω η συγγήτρια να απαντάει δημοσίως για το ποια θα είναι η διαπραγματευτική μας θέση. Γιατί, να υπενθυμίσω στην εισηγητρία, δεν χρειάζεται ε, το ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου για τις εξαιρέσεις αυτές, γιατί αυτή είναι η θέση που, στην οποία πρέπει να βασιστούμε. Κύριε Φέρμπερ, έχετε ερώτηση. Ναι. Ναι, δεκτό αυτό που λέτε. Αλλά πότε θα συζητηθεί το κάθε θέμα. Θα ήταν καλό να ξέρουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς την εισηγήτρια. Είναι εύκολη ερώτηση για τον επόμενο τριμερή διάλογο. Θα γίνει στον επόμενο τριμερή διάλογο, δηλαδή 10 Απριλίου. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Μετά την Κορεπέρ θα γίνει και γνωρίζουμε ότι γίνονται διάφορα παιχνίδια εκεί. 10 Απριλίου λοιπόν είναι ο επόμενος τριμερής διάλογος. Κύριε Πύρκε, κλείστε παρακαλώ το μικρόφωνο. Γιατί είστε πολύ ευηδείς, αλλά δεν χρειάζεται να σας έχουμε συνέχεια στην οθόνη. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ. Είχα πει και προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, αντίθετη στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της κοινωνικής νομοθεσίας. Ήταν κάθετα αντίθετη. Και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ε, οικοδομικών υλικών, τη μεταφορά των τούβλων. Και εκεί ήταν κατηγορηματική ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν κατά. Γιατί δηλαδή να είναι διαφορετική μεταφορά των τούβλων από την μεταφορά άλλων αγαθών ή τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ταχθεί κατά των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και κατά τις ταχυδρομικες υπηρεσιες η ευρωπαικη επιτροπη λοιπον ταχθηκε κατα των τροπολογιων του ευρωπαικου κοινοβουλιου ακομη και κατα τις τροπολογιες που ζητούσε 2,8 αντί για 3,5 τόνους. Η μοναδική εξαίρεση που προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε και που είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για να δεχτούμε την συμφωνία είναι η πανευρωπαϊκή εξαίρεση ε, στο άρθρο 3, δηλαδή μία ακτίνα 100 χιλιόμετρων από την έδρα της εταιρεία για, τα, για μη επαγγελματίες οδηγούς και για φορτηγά κάτω των 7,5 τόνων. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό γιατί μιλάμε για μη επαγγελματίες οδηγούς, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνουμε μάχη με νύχια και με δόντια για να διαφυλάξουμε αυτή την εξαίρεση. Άλλωστε είναι η μοναδική εξαίρεση ε, που δεν βρήκε απόλυτα κατηγορηματική και αντίθετη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και συνεχίζουμε το διάλογο και ευελπιστούμε ότι θα τη μεταπίσουμε τελικά. Όπως είπαμε, ο επόμενο τριμερή διάλογο θα γίνει στι 10 Απριλίου. Θα είμαι παρόν εκεί, όχι γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στην ε, ε, εισηγήτρια, αλίμονο, αλλά πιστεύω ότι καλό θα είναι να έχουμε, να έχουμε μια επίβλεψη να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και θα επανέλθουμε μετά τον τριμερή διάλογο και θα σας ενημερώσουμε για το τι συμφωνήθηκε, τι όχι και τότε ίσως γίνει συζήτηση. Για το ίδιο θέμα... Επειδή ακούστηκαν διάφορα σχόλια, ε, καλό είναι να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση για να παρέμβουμε και στις κυβερνήσεις μας, μήπως πετύχουμε τίποτα. Ναι. Μπορεί να σε σοκάρει αυτό το τζαζίν, αλλά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυρία Φώστερ έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή στην ε, κυβέρνηση από ότι εγώ. Αν εν πάση περιπτώσει, ε, το σχόλιο σας ε, το καταγράψαμε και ο κύριος Μπένιον το ίδιο. Πάμε στο δεύτερο τριμερή διάλογο, τέντη, κύριε Κουμουτσάκο, 20 Μαρτίου έγινε ο τριμερής διάλογος. Και μετά κύριος Χέρτοκ. Ε, δεν έχουμε λόγο, δεν βάλαμε την κυρία Γκουρμά για να τους χωρίσουμε, εξακολουθούν να έχουν θαυμάσει σχέση μεταξύ τους. Πρόεδρε, ο δεύτερος, ε, ο δεύτερος τρίλογος ε, μπορώ να πω ότι έγινε σε ένα πολύ καλό κλίμα και ήταν αποδοτικός. Είχε προηγηθεί ικανοποιητική προετοιμασία της συναντήσεως του Τριλόγου από τις τεχνικές επιτροπές, οι οποίες, θυμίζω, ε, είχαν με αποφασίσει στον πρώτο Τρίλογο να συσταθούν σε επίπεδο ε, συνεργατών και βοηθών, προκειμένου να ετοιμάζεται καλύτερα το έδαφος των Τριλόγων, πράγμα και το οποίο έγινε. Στον Τρίλογο αυτό συζητήθηκαν τρία βασικά τμήματα του ε, εγγράφου των κατευθυντηρίων γραμμών. Τα παραρτήματα, δηλαδή οι χάρτες, το κεφάλαιο 4 που αφορά τους διαδρόμους και τους συντονιστές και το κεφάλαιο 1 που αφορά το σύνολο των ορισμών, definitions, ε, των θεμελιωδών εκείνων ορισμών ε, που χρησιμοποιούμε στο κείμενο και είναι μεγάλης σημασίας για την ισορροπία και τη λογική του κειμένου. Το γενικό συμπέρασμα από τον δεύτερο τρίλογο είναι ότι το Συμβούλιο προσέρχεται με επικοδομητική διάθεση. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 4 που αναφέρεται στους διαδρόμους και τους συντονιστές, όπως θα σας πει σε λεπτομέρειες ο συνάδελφός μου κύριος Ερτούγκ, το Συμβούλιο έχει αποδεχθεί να καλύψει σημαντική απόσταση για να συναντήσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως η απόσταση παραμένει, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην καταγράψει την βούληση του Συμβουλίου να καλύψει επικοδομητικά μεγάλο μέρος της απόστασης ε, που χωρίζει τις θέσεις των δύο θεσμών. Το δεύτερο θετικό είναι ότι το Συμβούλιο αποδέχεται τις ε, implementing acts. Κάτι το οποίο και για μας αλλά και για την Επιτροπή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Βεβαίως, αυτές τις δύο θετικές στάσεις του και στο κεφάλαιο 4 και στο θέμα των Implementing Acts το Συμβούλιο τη συνδέει και απαιτεί μια μεγαλύτερη ευελιξία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύο πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέματα. Το ένα είναι το ζήτημα της, ε, της δέσμευσης χρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη. Είναι το σημείο 1-4 του κειμένου, αυτό που λέμε financial reserve, όπου θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και άρα ρηγότερη δέσμευση για την χρηματοδότηση των ε, σχεδίων που θα έχουν εγκριθεί. Και το δεύτερο, από το οποίο ζητάνε μεγαλύτερη ευελιξία από το ε, Κοινοβούλιο, αφορά τους χρονικούς, τα χρονικά όρια του 2030 και του 2050. Γιατί το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει δεδομένων των συνθήκων και των οικονομικών ευρύτερα αλλά και επιμέρους επιχειρημάτων που παρουσίασαν ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία. Και στα δύο αυτά ζητήματα, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σεβόμενη την εντολή που έχουμε, δεν ε, πήραμε καμία δέσμευση και δεν αποδεχθήκαμε τη λογική που ε, θέλει το Συμβούλιο. Ειδικά τονίσαμε ότι το χρονικό όριο του 2030 για το Core Network είναι μη διαπραγματεύσιμο. Για το 2050 επίσης τονίσαμε την βούληση του Κοινοβουλίου να παραμείνει ως έχει και σε περίπτωση, επειδή πραγματικά είναι ένα χρονικό όριο που είναι μακριά στο μέλλον, θα χρειαστεί κάποια ευελιξία, αυτό από πλευράς μας θα συνδεθεί και θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και στα άλλα σημαντικά κεφάλαια του εγγράφου. Δηλαδή τα κεφάλαια 2 και 3 που αφορούν τα technical requirements και άλλα. Ε, κλείνοντας αυτή την εισαγωγική ε, παρέμβαση, θέλω να συγκρατήσετε ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κινείται σε αρκετά σημεία του κειμένου σε μια κατεύθυνση να συναντήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό συνδέεται από πλευράς τους με αιτήματα ε, δικής μας σε ζητήματα τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί θεμελιώδου σημασία και θα διαπραγματευτεί πολύ σκληρά μέχρι το τέλο στο πλαίσιο τη εντολή που έχουμε πάρει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε έχετε να κάτι. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σε κάποιες λεπτομερείς για να ξέρουμε και τι συζητάμε. Ο κύριος Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 και τους διαδρόμους. Ένα βασικό κομμάτι όλης αυτής της ε, νομοθεσίας. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία στον τριμερή διάλογο, αλλά υπάρχουν και διαφορές που βρίσκονται ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 4. Εδώ πέρα θέλουμε ως Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την έντολή μας, να επιμείνουμε στη δομή των διαδρόμων και στις πλατφόρμες των διαδρόμων. Οι συντονιστές των διαδρόμων πρέπει να έχουν και σαφείς ε, αρμοδιότητες για όλους ε, για όλες αυτές τις περιπτώσεις και το ERTMS και τους, ε, τις λεωφόρους της θάλασσας. Και βεβαίως πρέπει εδώ πέρα να συμπεριληφθούν επαρκώς, ε, να συμπεριληφθεί το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εδώ πέρα φέρνει αντιρρήσεις στο Συμβούλιο, αλλά ελπίζουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο να καταλήξουμε σε κάποια διατύπωση. Σε αυτά τα τρία σημεία όμως νομίζω πως μπορούμε να είμαστε επιτυχείς ε, Την τελευταία εβδομάδα ε, ενημερωθήκαμε πως υπάρχουν διαφορές για το πώς ε, θα πρέπει να είναι αυτή η πλατφόρμα του διαδρόμων. Το Συμβούλιο μίλησε για κάποιες ομάδες εργασίας ad hoc. Τελικά συνεννοηθήκαμε σε ένα σταθερό μοντέλο των φόρουμ των ε, διαδρόμων και αυτό βεβαίως σε συνεργασία με τους συντονιστές. Όσον αφορά λοιπόν τον ρόλο των συντονιστών μπορούμε νομίζω να συμφωνήσουμε στι, στις αποστολές που θα έχουν ε, και για το ERTMS και για τις ε, λεωφόρους θάλασσας. Ο συμβασμός λοιπόν αυτός είναι ένα πρώτο βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά εδώ πέρα, ε, όπως είπαμε, υπάρχει σαφώς ε, η ανάγκη βελτίωσης. Βεβαίως κάτι άλλο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι η ευθυγράμμιση, ο συγχρονισμός, εάν θέλετε, των ε, διαδρόμων αυτών για το σιδηροδρομικό, για τις εμπορευματικές μεταφορές με τον ε, σιδηρόδρομο. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να είμαστε αρκετά ευέλικτοι και να μην δημιουργήσουμε διπλές δομές, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει μια ε, κάποια λειτουργικότητα. Όσον αφορά το κεφάλαιο 1, αναφέρθηκε πως ε, τα δύσκολα ζητήματα είναι στο άρθρο 1 παράγραφος 4 για τις προθεσμίες και τη δεσμευτικότητα. Καταλαβαίνετε πως εδώ πέρα το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να το νερώσει λίγο αυτό, αλλά δεν συμφωνούμε βεβαίως και ως Κοινοβούλιο έχουμε μια ξεκαθαρή θέση. Δηλαδή, να μην επιτρέψουμε ε, κάποιες ε, προθεσμίες ε, για την ε, χρηματοδότηση και το 2013 και 2015. Αλλά σωστά είπε ο κ. Κουμτσάκος πως ε, όταν έχουμε ένα μακροπρόθεσμο διάστημα μέχρι το, 2010, μέχρι το 2050 ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Ε, Επίση, αυτό το οποίο είναι σημαντικό με τους ορισμούς στο κεφάλαιο 1 είναι σημαντικό να ορίσουμε και την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να α, συμφωνήσουμε Συμβούλιο και Κοινοβουλίο. Εντάξει, εδώ πέρα υπήρξε κάποια μετακίνηση, αλλά θα πρέπει να τα δούμε αυτά με την... μέχρι την άλλη φορά. Και επίσης μια μεγάλη επιτυχία είναι το Συμβούλιο διατεθειμένο να προσθέσουμε έναν ορισμό για την ε, κοινωνικο-οικονομική μελέτη επιπτώσεων και για το κλίμα. Κάτι στο οποίο επέμενε το Κοινοβούλιο. Και τέλος, καταφέραμε ως ε, Κοινοβούλιο να ε, προχωρήσουμε στις, ε, στην κατηγοριοποίησή μας για τους στόχους, την συνοχή, τους χρήστες και νομίζω πως θα προσπαθήσουμε και το διάστημα που έρχεται να έχουμε μια κοινή προσέγγιση με το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη όσον αφορά τους ορισμούς. Νομίζω πως θα το πετύχουμε. Αυτό νομίζω το δέχεται και η Κομισιόν και το Συμβουλίο. Αυτά και ο επόμενος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα 25 Απριλίου. Σας ευχαριστώ. Ξεκινήσουμε τον κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων. Να σα επενθυμίσω ότι πρόκειται περί ε, ενημερώσεω όσον αφορά το όλο θέμα. Δεν πρόκειται για νέα συζήτηση. Και κάποια πράγματα ίσω δεν πρέπει να τα συζητάμε δημοσίω μέχρι ότου να είμαστε σε μια θέση για να τα πραγματευτούμε. Γιατί και τύχη έχουν αυτοί, όπω λένε. Ξέρετε, ε, υποτίθεται ότι πρέπει να συμμορφωθούμε το άρθρο 17, πρέπει να είναι μια σύντομη ενημέρωση τώρα, αν και να δούμε αν υπάρχουν ερω... σύντομε ερωτήσει και να το έχει υπόψη η συγγήτρια για το μέλλον. Έχουμε με χρόνο μεν σήμερα. Σα διαβεβαιώ όμω ότι όταν μπούμε στο πακέτο για του σιδηροδρόμου και άλλα μεγάλα θέματα που θα συζητήσουμε, δεν θα έχουμε χρόνο, ούτω ώστε κάθε συγγητή να μιλάει για 10 λεπτά και να αναφέρεται στα τεκτενόμενα στου τριμερείς διαλόγους. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ο κύριο Πέρκερ, μπορεί να υποβάλουν ερωτήσει. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποιε ερωτήσει. Πάντω με καθησύχασαν οι δύο εισηγητέ, γιατί η ελαστικότητα που ζητά το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη σύνδεση τη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη δεν είναι δυνατή. Είναι ένα από τα καινοτόμα σημεία αυτής της προσπάθειας, ούτε έχουμε ελαστικοποίηση των ε, χρονικών ορίων. Γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα χρονικά όρια για να αποκλειστούν κάποιες σημαντικές υποδομές. Οπότε, αν έχουμε ευελιξία σε αυτό το θέμα, επαναρχόμαστε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη προσπάθεια. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ερτούκ, να εμείνουμε στη θέση μας, γιατί αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του, της νέας μας προσπάθειας. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις. Το συζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ευθυγραμμίσει τον κανονισμό για τα εμπορεύματα, τα, τους διαδρόμους εμπορευμάτων. Ήταν θέμα διαχείρισης, συμφωνιών διαχείρισης για διάφορους διαδρόμους, για υπάρχουσες υφιστάμενες υποδομές με τον ισχύοντα κανονισμό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι καταλάβαμε προσπαθεί να τροποποιήσει τον κανονισμό για τους διαδρόμους εμπορευμάτων που ήταν ε, κανονισμός που αφορούσε οι υφιστάμενες υποδομές και τους, ε, τη χαρτογράφηση και τη χρηματοδότηση των ε, διαδρόμων του ΣΕΦ. Ο διάδρομος από το Ταλίν στην Βενετία κονα θα έκανε μία παρέκκληση από Βαρσοβία και θα οδηγούσε στο Ρότερνταμ. Ερωτήσεις παρακαλώ, ερωτήσεις θέλουμε εδώ, όχι παρατηρήσεις. Μα ερώτηση υποβάλλω. Μα θέστε την ερώτηση επιτέλους. Ερώτηση. Μα δεν εξηγήσω. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ε, ξανα... Συζητάμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Γνωρίζουμε τι συμφωνήσαμε, έχουμε πρώτη ανάγνωση, γνωρίζουμε τη, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτά τα ξέρουμε. Η ενημέρωση έγινε για τις διαπραγματεύσεις, από την έκβαση του πρώτου τριμερούς διαλόγου. Αυτό που περιμένουμε από τα μέλη τώρα είναι να υποβάλουν ερωτήσεις ή απορίες τους προς τους συγκητές για αυτά που είπαν. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε συζήτηση για το τι είναι η διάδρομη εμπορευμάτων. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Μόνο ερωτήσεις, ερωτήσεις και απορίες. Με αυτό ρωτάω κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα TENS που επηρεάζει και τη ΣΕΦ. Είναι κάτι καινούριο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και ρωτώ του συναδέλφου που δεν το ανέφεραν προηγουμένω. Αυτό το σημείο συζητήθηκε. Είναι κάτι καινούριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με και τους δύο κανονισμούς. Γίνεται μια ευθυγράμμιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Συζητήθηκε αυτό. Δεν προσπαθώ να κάνω συζήτηση. Θεωρώ, ε, για τι έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση κάποιε προσθήκε που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε ότι 38 λιμάνια ε, ποταμών ε, ζητήθηκαν από την γερμανική κυβέρνηση. Θα συζητηθεί αυτό, θα τροποποιηθεί κάτι από αυτά που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρωτά λοιπόν για τις αλλαγές κύριε Πρόεδρε, να δω τι αλλαγές έγιναν στις διαπραγματεύσεις, γιατί επηρεάζουν το ΣΕΦ το Connecting Europe Facility. Γι' αυτό έθεσα τις ερωτήσεις. Κύριε Πέρκερ, δεν υπάρχουν αλλαγές. Κανείς δεν πρότεινε ακόμα αλλαγές. Ο κύριος Πέρκερ έχει το λόγο. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι συντονιστές αναφέρθηκαν σε ένα βασικό δίκτυο το οποίο έγινε σωστά, αν κατάλαβα καλά. Ο κύριος Ερτούγ είπε πως υπάρχουν διαφορές. Το ερώτημά μου είναι γίνεται δεκτό πώς θα υπάρξουν οι δέκα βασικοί διάδρομοι που έχουμε προτείνει. Δεύτερο ερώτημα προς συντονιστές. Ε, αυτοί έγιναν δεκτοί, αλλά το θέμα είναι έγινε δεκτός και ο μηχανισμός ελέγχου που προβλέπουμε και αυτά τα οποία εμείς ε, προβλέπουμε ως συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης ε, διατάξεων κτλ. από την Κομισιόν. Κύριε Γκρός. Απλή ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Αυτό αφορά και τις δύο εκθέσεις. Πάντα αναζητούσαμε μία συνέπεια μεταξύ των διαδρόμων και του Μεσοσυνδέτα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μάθω αυτή τη στιγμή πώς θα διασφαλιστεί αυτή η συνέπεια στον ε, τριμερή διάλογο. Κύριε Ρίκη. Σύντομη ερώτηση. Άκουσα τον Γιώργο να μιλήσει για εκτελεστικές πράξεις. Υπήρξε κάποια πρόοδος, κάποια πρόταση του Συμβουλίου όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των κατοξισουδότησης πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Από τους συζητητές ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Γιώργο. για το ερώτημα του κυρίου Ερικέ. Πρόεδρε, έκανα εγώ λάθος. Εγώ αναφέρθηκα στην παρέμβασή μου στο ότι συζητήσαμε και τα παρατήματα τους χάρτες και δεν είπα τίποτα πάνω σε αυτό, σχεδόν τίποτα. Τώρα έχω τη δυνατότητα να σας ε, δώσω μια γενική ιδέα της πορείας των συζητήσεων για τα παρατήματα και για τους χάρτες. Και τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν προκατακτικά να κλείσει το κεφάλαιο ε, για, για τους χάρτες. Αποτελείται το κεφάλαιο από τις τροπολογίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύο επεξηγηματικά έγγραφα συμπεριλαμβάνονται που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας είπε σαφώς ότι όλες αυτές οι αλλαγές ευθυγραμμίζονται με τη μεθοδολογία και τα δύο θεσμικά όργανα μπορούν καταρχήν να αποδεχθούν σχεδόν όλες αυτές τις αλλαγές, κάποιες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, όμως δεν έγιναν ακόμα δεκτές από το Συμβούλιο. Και βέβαια, εμείς επιμένουμε στις θέσεις μας. Άλλη εκκρεμότητα, το δεύτερο σημείο που αφορά τα παρατήματα, και εκρεμή αφορά τις αλλαγές αυτές που περιστρέφονται γύρω από την προσχώρηση της Κροατίας. Αυτά είναι κρεμή ζητήματα. Προσωρινά σταμάτησε η συζήτηση για τους χάρτες, διότι πρέπει να γίνουν πολλά στους επόμενους τριμερείς διαλόγους. Αυτή είναι, αυτό εννοείται. Όσον αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις, πράγματι το Συμβούλιο είπε ότι μπορεί να συμφωνήσει και μπορεί να τις δεχτεί. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Χέτσογκ, να έχετε κάτι να προσθέσετε. Ε, Ευχαριστώ και για όσους ε, έκανα. Ευχαριστώ όσους έκανα ερωτήσεις. Τώρα για το έρθμα της κυρίας Αγιάλα Σέντερ για τους ε, διαδρόμους. Η προσέγγιση μας είναι πως βεβαίως εκπροσωπούμε την άποψη του Κοινοβουλίου. Και βεβαίω προσπαθούμε να επιτύχουμε δύο στόχου. Πρώτον, να μην έχουμε διπλέ δομέ και δεύτερον, να υπάρχει λειτουργικότητα. Και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια πρόταση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση το πώ σκοπεύει να επιτύχει αυτούς τους δύο στόχους. Για το θέμα του κυρίου Γκρός, για το πώς ε, θα επιτευχθεί αυτή η συνέπεια και με το μέσο συνέδρας ε, την Ευρώπη. Βεβαίω αυτό είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικό και, και η γραμματεία μας βεβαίω ε, το προσέχει έτσι ώστε οι ορισμοί να είναι οι ίδιοι και το υπενθυμίσαμε και στον τριμερή διάλογο. Δηλαδή όταν κάτι δεν ήταν σαφές το αφήνουμε κατά μέρο, ε, γίνεται μια συνεννόηση μεταξύ των δύο εισηγητών και μετά συζητάμε το Συμβούλιο. Μη φοβάστε. Ε, και μόνοι μας το φροντίζουμε αυτό. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται δύσκολο όταν έχουμε 4-6 εισηγητέ, αλλά προσπαθούμε και βεβαίω ε, είναι και στι δύο διαβουλεύσει η βοηθή μα. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Πίρκερ για το αν γίνεται αποτεκτό το βασικό δίκτυο. Το Συμβούλιο δέχτηκε πράγματι την ε, διτή αυτή προσέγγιση και για τον μηχανισμό ελέγχου είπα πως δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει εδώ πέρα. Το κοινοβούλιο, το συμβούλιο μου συγχωρείτε, έρχεται πιο πολύ προς το ε, Προ τι δικέ μα θέσει για το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι πλατφόρμες, ή φόρουμ των διαδρόμων. Οπότε μέχρι την επόμενη συνάντηση νομίζω θα έχουμε καταλήξει κάτι και αυτό βέβαια και πηγαίνει προ την κατεύθυνση αυτού του οποίου είπε ο κ. Κουμουτσάκο. Είμαστε πολύ προσεκτικοί ως ε, Κοινοβούλιο για το τι αρμοδιότητες δίνουμε στην Κομισιόν. Απλά στην περίπτωση αυτή είναι σωστό νομίζουμε και η Κομισιόν να γνωρίζει εδώ πέρα το τι θα γίνει. Για τους διαδρόμους λοιπόν μην ε, ανησυχείτε, θα, θα δώσουμε βάρος και στην επόμενη τριμμένη. Συνάδελφοι, Μάικλ, κοίτα, ανησυχώ διότι το Συμβούλιο ποτέ, ποτέ μα ποτέ των ποτών δεν συζητά δημοσία τα όσα συμβαίνουν εκεί. Και εδώ είμαστε ανοιχτοί όσο πιο πολύ συζητούμε, τόσο πιο πολύ προδίδουμε τις θέσεις μας. Και γι' αυτό δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να σας το πω, Μάικλ. Μα ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να πω κάτι. Όλα αυτά ακούγονται θαυμάσια, ότι πηγαίνουν θαυμάσια και τα βασικά σημεία δεν είναι καν στη μερίσια διάταξη και δεν έχουμε συμφωνήσει. Αν σκεφτείτε ε, πως ε, το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ... Άμα λέτε δηλαδή εδώ μέσα πως το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ προσιτό κτλ. Ε, δεν είναι δυνατό να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα δημοσίως. Ε, αυτά έπρεπε να τα συζητάμε και κλεισμένων των θυρών. Τη δε Κομισιόν θα έπρεπε να μας έχει στείλει τον ε, κατάλογο για τους διαδρόμους, δεν τον έχουμε ακόμα. Δεύτερον, τα λεφτά. Πού θα τα βρούμε. Δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε μια θαυμάσια λίστα. Έχει τους λόγους του βεβαίω το Συμβούλιο, ούτε αυτό το έχουμε συζητήσει. Τα δύσκολα λοιπόν θα έρθουν. Οπότε αν δημιουργείται εδώ πέρα η εντύπωση πως όλα πηγαίνουν θαυμάσια με το Συμβούλιο, προσέξτε πάρα πολύ. Στα μικρά θα ε, συμφωνήσουμε. Τα μεγάλα έχουν αναβληθεί και αυτή η συζήτηση οπωσδήποτε δεν πρέπει να γίνεται δημόσια. Είμαι πολύ δυσαρεστημένος από την πορεία. Γιώργο να μιλήσεις, αλλά παρακαλώ. Δεν είμαστε εδώ για μια ανοιχτή συζήτηση. Ας στείλουμε και στο Συμβούλιο ένα γράμμα. Γιώργο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Και εντάξει, έχω επίγνωση των όσων λέτε και θα είμαι προσεκτικό. και προσπάθησα να είμαι προσεκτικό στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Αναφέρθηκα σε μια θετική ατμόσφαιρα στην περασμένη συνεδρίαση. Αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο απεδέχθη τα πάντα που επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Ήταν η ατμόσφαιρα που κράτησε μια συνάντηση και είπα ότι το βασικό κομμάτι, το σημαντικότερο του εγγράφου παραμένει ανοιχτό και θα παραμείνουμε στα πλαίσια τη δολή που μα ανατέθηκε. Αυτή είναι η κατάσταση. Το να πω κάτι διαφορετικό θα ήταν εσφαλμένο. Πρόεδρος, θα προχωρήσουμε. Ε, ε, έτσι γίνεται. Άμα ξεκινήσει, ε, ανοίγει συζήτηση. Δεν θέλω κάτι τέτοιο. Στι σημειώσει μου εδώ λέει, υπενθυμίσα στα μέλη ότι πρόκειται περί τυπική διαδικασία και δεν θα πρέπει να ανοίξει ουσιαστική συζήτηση. Απέτυχα παταγωδό αυτό και παραδέχομαι την ενοχή μου. Εδώ πρόκειται περί ενημέρωσης. Μία ενημέρωση. Όχι να τους δώσουμε αυτό, να τους δώσουμε το άλλο, γιατί δεν κάνουμε το ένα, γιατί δεν κάνουμε το άλλο. Ενημέρωση, σας παρακαλώ. Τι απέρευσε από όλα αυτά. Σύμφωνα με το άρθρο 70 πρέπει να πάμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Το άρθρο 70 υπονομεύει τελικά τη θέση του Κοινοβουλίου. Αν πρέπει να το κάνουμε αυτό δημοσία, όπως σωστά είπε και ο Μάικλ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο ΣΕΦ, στο επόμενο θέμα, στον κύριο Ρίκε, κυρία Αγιάλα Σέντερ. Και στις σημειώσεις μου λέει ότι είναι μια διαδικασία και δεν θα ανοίξει επί της ουσίας η συζήτηση. Ο κύριος ε, Ρίκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα έγινε ο πρώτος τιμής διάλογος όσον αφορά το Connecting Europe Facility και αναφερθήκαμε στα βασικά σημεία που αποτελούσαν αντικείμενο αποκλήσεων. Και θα ήθελα να παραθέσω εντάχυτα σε σημεία αυτά, τα αριθμητικά στοιχεία, διότι πρόκειται περί χρηματοστικού εργαλείου και αυτά συζητούνται στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, η εισαγωγή του, της ευελιξίας, η χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων, που το Συμβούλιο διστάζει πολύ πάνω σε αυτά από τι κατεξουδότηση πράξει να περάσουμε σε εκτελεστικέ πράξει. Προασπίζεται το Κοινοβούλιο προφανώ τι κατεξουδότηση πράξει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι εκτελεστικέ. Ευθυγράμμιση των παρατημάτων είναι κάτι που αναφέρθηκε και μετά κάποιοι κανόνες, μηνότητες, υπάρχουν διαφορέ, εισαγωγή ε, του ΦΠΑ, παραδείγματο χάρη, χρηματοδότηση ε, τα δίχτυα που συμπεριλαμβάνονται, διάφοροι, διάφορες διαδρομές και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι κάποιες δυσκολίες δεν μας επηρεάζουν εμάς αλλά θα επηρεάσουν τη Γενική Συμφωνία όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια όπου υπάρχει άρνηση του Συμβουλίου να λάβει υπόψη ότι αυτά που έχουν ληφθεί στο, υπόψη στο παράρτημα, στο, στα παρατήματα του ΣΕΦ θέλουν αυτοί μάλλον να καθορίσουν τις καθεδίες γραμμές για την ενέργεια. Όλα αυτά θα υπονομεύσουν σοβαρά τη γενική συζήτηση για το μέσο αυτό του το Connecting Europe Facility, το SEF. Αυτά κάναμε στον πρώτο τιμερή διάλογο. Εξετάσαμε όλα αυτά, δηλαδή τα σημεία που δημιουργούσε συζήτηση, που δεν πήγαν καλά. Το πνεύμα συνεργασίας ήταν εξαίρετο, διότι δεν αντιμετωπίσαμε τα σημεία εκείνα που θα μπορούσαν επίμαχα. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο Ντομινίκ Ρικέ και να προσθέσω ότι επιμείναμε πολύ στο θέμα της χρηματοδότησης. Απαιτήσαμε από την, Ευρω... από την Ελλανδική Προεδρία να μας ενημερώσει, να μας πει τι γίνεται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αντιστάθηκε, εμείς επιμείναμε και είπαμε ότι δεν μπορούν όλα να μας τα επιβάλλει το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και εμείς ως ε, ε, ε, διευκόλυνση ιδέων στην Ευρώπη έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε για την εσωτερική κατανομή των κονδύλιων. Επίσης, μιλήσαμε για το θέμα της εναρμόνισης, όπως είπε ο κ. Κρόης, μεταξύ των δύο κανονισμών του ΣΕΦ, του Connecting Europe Facility και των κατευθυντηρίων γραμμών. Και όπως είπε ο κ. πρέπει να προσέξουμε το θέμα των ορισμών. Για γι' αυτό θα γίνει κοινή συνεδρίαση, για να ε, πραγματώσουμε αυτή την εναρμόνιση. Υπάρχουν ερωτήσεις για το Connecting Europe Facility, το ΣΕΦ. Όχι. Mr. Ferber. Ο κύριος Φέρμπερ. Ε, τα ενδοκοινοβουλευτικά θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τη steering group και με το δημοσιονομικό πλαίσιο του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν γίνεται οι να λένε θέλουμε περισσότερα λεφτά και οι δε να λένε δεν υπάρχουν. Τι διαδικασία προβλέπετε λοιπόν. Well, Είμαι σε αυτή την επιτροπή και η περιγραφή σας ήταν άριστη κύριε Φέρμπερ επίκειται κάποια συνεδρίαση μετά το Πάσχα. Δεν μπορώ να παραστώ. Θα ζητήσω τον Ντομινίκ να παραστεί. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια δηλαδή. Σεφ και αντιπρόεδρος. Ποια είναι η εντύπωσή μου. Γίνονται αυτές οι συναντήσεις οι ανωτέρες δυνάμεις παίρνουν τις αποφάσεις, αν το πω διπλωματικά. Έχω προβλήματα και από εθνική σκοπιά εγώ. Ο πρόεδρος προωθεί τις υποθέσεις μαζί με τον κύριο Λαμασούρ, κύριο Γκάλφιν, κύριο Σμπόγκε. κάνουν τα δικά τους και οι υπόλοιποι εμείς είμαστε απλώς θεατές μερικές φορές. Πολεμούν όλοι για τη θέση στην Επιτροπή, ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό. Σύντομα. Είναι. Και εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή. Είμαι αρμόδια για τον κανονισμό το Connecting, Connecting Europe Facility και υπενθυμίζουμε ότι η κατανομή, υποδομές και η ανανέωση των υποδομών, ο ξεχρονισμός του είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να εξασφαλιστεί η δέουσα χρηματοδότηση αυτής της διευκόλυνσης. Ο Ντομινίκ, ευχαριστώ. Εγώ είμαι ο εισηγητής της ομάδας μας για τον προπολογισμό του 2014 και μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής μας προσπίζουμε τα συμφέροντα της Επιτροπής Μεταφορών στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Έχουμε μια ομάδα επαφής. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Επόμενο σημείο είναι το εργαστήριο ενημέρωση επισκόπηση των συμφωνιών που έχουν συναυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των υπηρεσιών, των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Είναι εδώ οι ομιλητές, θα ξεκινήσουμε ένα πεντάλεπτο για να οργανωθούμε. Λοιπόν, στις και 20, πέντε λεπτά διάλειμμα για ένα καφεδάκι. Colleagues, can I ask you to take your seats again, please? Next item on the agenda. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη Έχουμε επισκόπηση των συμφωνιών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών που έχουν συναυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις φιλοξενούμες θα κάνουν παρουσιάσει εδώ. Ο κύριος Εβεν Κβαντεστάινεν, Κλοντ Πρόπστ και Χουσίν Κάν τρεις καλεσμένοι. Με αυτή τη σειρά θα μιλήσουν, αν συμφωνούν όλοι. Με αυτή τη σειρά τους παρουσιάζω. Καλώς. Θα μας σχολιάσουν την όλη κατάσταση πριν σας δώσω το λόγο. Έχουμε λοιπόν την ε, αναφορά, την έκθεση αυτή εδώ. Έχουμε τους εμπειρογνώμονες. Θα ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να μιλήσουν ο καθένας για ένα δεκάλεπτο. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Βόντενστάινεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Καλημέρα να πω όλους, μη και ξεκινάω εγώ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εμφανιστώ εδώ. Μετά από εισαγωγικά σχόλια θα αναφερθώ λοιπόν στο θέμα των συμφωνιών. Ε, υπάρχει συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και συμφωνία με τον Καναδά, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα με ακούτε τώρα. Ξεκινώντας έχω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά τους τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα όλοι οι πυλώνες αντικατοπτρίζουν στρατηγική για ανοιχτό και θεμητό ανταγωνισμό στις διεθνείς αερομεταφορές και τις σχετικές αγορές. Και συμφωνίες του πυλώνα 1 που επιβάλλουν αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης διμερείς ε, έχουν, ε, αφορούν την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά οι διαπραγματεύσει πυλώνα 2 και πυλώνα 3 με εταίρου εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι να επιβάλλουν στο βαθμό του δυνατού τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω Συμφωνία και, και εταίρο τρίτου πυλώνα εξαρτάται από τρία κριτήρια, δύο κριτήρια μάλλον. Πρώτα απ' όλα η οικονομική συμφων... σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η συμφωνία και δεύτερον η πολιτική προθυμία να υπάρχουν κοινοί ρυθμιστικοί στόχοι που θα επιδιώκονται. Οι μικρότερες αγορές εξακολουθούν να ρυθμίζονται αποτελεσματικά σε επίπεδο κρατών μελών κυρίως όταν οι εφικτές διαδρομές ε, αφορούν ένα ή εμπλέκουν ένα ή δύο και όχι περισσότερα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις πυλώνα 3 με τη ΣΥΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά. Λοιπόν, καταλήξαμε σε συμφωνίες ανοιχτές των αερομεταφορών. Και όσο εκτελήσονται οι διαπραγματεύσει, ακολούθησαν δύο διαδρομέ συζητήσει. Πρώτα απ' όλα, απελευθέρωση των αγορών, που σημαίνει άρση ποσοτικών ελέγχων όσον αφορά τη δυναμικότητα και τις τιμές των διαδρομών και ρυθμιστική σύγκληση από την άλλη, που σημαίνει την επιβολή κοινών προδιαγραφών όσον αφορά τη θέτηση θεμάτων ασφαλείας, ε, περιβάλλοντος, ε, θεμητού ανταγωνισμού, ε, σωστών συνθήκων εργασίας και ασφαλείας των αερογραμμών. Λοιπόν, η επελευθέρωση και η απορρίθμιση σημαίνει οι κανόνες να φεύγουν ε, αφορούν σχέση ενός με κάποιον άλλον. Και έτσι γίνεται μια ομαλοποίηση των διαδρομών. Είναι λογικό αυτό όπω γίνεται στην ΕΠΑ. Αν πιστεύει κανεί ότι πραγματικά η ελευθερία ανταγωνισμού απαιτεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, η απελευθέρωση θεωρείται σαν λογική συνέπεια της σύγκλησης, τη δομή, ισότιμη αντιμετώπιση υπό ίσε συνθήκε. Στην όλη δομή εδώ ε, έχουμε διαφορετικέ συμφωνίε από ό,τι κατά το παρελθόν όσον αφορά το φάσμα των καλυμμένων θεμάτων και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, όπω να υπάρχει μια μεικτή επιτροπή Λοιπόν, ορισμού αυτές οι συμφωνίες συνεπάγονται ε, να δημιουργείται ένας χώρος, ένα περιφερεια, μια περιφερειακή αγορά και ένα πλαίσιο. Προς, με, ακολουθήσαμε τις μετεθμίσεις ε, που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών προς τις τρίτες χώρες. Θέλουμε όμως αυτές οι συμφωνίες να είναι κάτι παραπάνω παρά γεφύρωση μεταξύ διαφόρων ρυθμισμένων εθνικών αγορών. Και τέλο, να πω κάτι για την διαδικασία και πώ ακολουθούνται διάφορα στέδια. Προσέγγιση που ακολουθείται στι διαπραγματεύσει του πυλώνα 3 και σε κάποιε περιπτώσει του πυλώνα 2. Δηλαδή, βήμα-βήμα προχωράμε. Είναι λογική η μέθοδο αυτή για μια φιλόδοξη προσέγγιση, αλλά χρειάζεται να καθορίσει κάποιε φάσει με ρεαλιστικό τρόπο Τώρα πάμε στη Συμφωνία ΕΕ Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ξεκινάμε με το πριν και μετά, σύγκριση πριν και μετά. Τι άλλαξε εν συγκρίση με το status quo που, εκ των προτέρων, που ίσχυε πρωτήτερα. Με τη ΣΥΠΑ τα κράτη-μέλη αντιμετώπιζαν έναν εταίρο που ακολουθούσε συνεπείς πολιτικές όταν ε, να διαπραγματεύσεις με την Ολλανδία το 1992 για ανοιχτούς ουρανούς. Αυτή η συμφωνία ήρε όλους τους περιορισμούς όσον αφορά τις κλασικές διαδρομές και άνοιξαν και δυνατότητες να συνεργάζονται αεροπορικές εταιρείες και να δημιουργούν δίκτυα και να ωφελούν έτσι τους καταναλωτές. Τα χρόνια που ακολούθησαν, τα περισσότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω διαπραγματεύτηκαν ουσιαστικά ταυτόσιμε παρόμοιε ρυθμίσει με τη ΣΥΠΑ. Βασική εξαίρεση ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο που επέμεινε επί βαθύτερη δίζηση τη αγορά μέσω επενδυτικών δικαιωμάτων σε αντάλλαγμα αποδοχή αμερικανικού τύπου απελευθερώσεων των αγορών όταν δεν επετέφθησαν αυτέ τα διαπραγματευτικά δικαιώματα οδηγήθηκε οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα μπλεκόμενοι ότι αυτή η συμφωνία δεν προσέθεται πολλά ωφελήματα για την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Η νέα συμφωνία όμω πέτυχε κάποια νέα δικαιώματα για του μεταφορέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ανοίχθηκαν 7η ελευθερία για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Οι ανταγωνιστέ των ΗΠΑ δεν πήραν κάτι καινούριο, εκτό εάν απελευθερωθούν τα επενδυτικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήθελε να απελευθερώσει τι επενδύσει, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει το Κογκρέσο να χαλαρώσει την νομοθεσία όσο δεν δίνονται επενδυτικά δικαιώματα, συμφώνησαν όμως οι ΙΠΑ τρίτη, μεταφορείς τρίτων χωρών που υπό την διοκτησία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να έχουν αυτή την πρόσβαση. Και απεδέχθηκε, απεδέχθηκαν οι ΙΠΑ διάφορε απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και υπήρξε ασφάλεια δικαιώσεων όσον αφορά επενδύσει διασυνοριακέ. Τέλο, οι ΗΠΑ δέχτηκαν διαδικαστικέ καινοτομίε όπω μια μεικτή επιτροπή και ε, είναι μια θεσμική μορφή που πριν δεν είχε γίνει αποδεκτή σε αρμοτεφορές. Πόσο συμφωνία είναι, θα είναι αυτή η μεικτή επιτροπή Ένωση, όπω είπα, θα το δούμε. Ένα τέτοιο μηχανισμό είναι κάτι σχετικό ως εργαλείο για βέλτιστη χρήση καθορισμό ε, μηχανισμών και να είναι και αποδοτικά τα μέτρα που εφαρμόζονται. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αγορά μεταφορών στον κόσμο να συνεχίζουμε να, μέσω, σε επίπεδο διμερών συμφωνιών 100 μελών να πετύχουμε μια συμφωνία στον τομέα θα ήταν κάτι επιστοδρομικό. Στο έγγραφό μου αναφέρονται κάποιε λεπτομέρειε στην περίπλοκη συμφωνία, αλλά θέλω να περάσω τώρα στον Καναδά, όπου αυτή η συμφωνία έχει ομοιότητε και σημαντικέ διαφορέ όσον αφορά την προηγούμενη συμφωνία που ανέφερα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτειών. Στην περίπτωση του Καναδά, το status quo ante είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Το 1 τρίτο των 100 μελών δεν είχαν καμία συμφωνία. Οι συμφωνίες των 18 που είχαν συναυθεί ήταν εμβαλωματικές. Αφορούσαν τα δικαιώματα. Λοιπόν, τρεις ήταν φιλελεύθερες, δύο με τέσσερις συμφωνίες ήταν με τρίους ανοιχτές όσον αφορά στην αγορά και τις σχετικές ελευθερίες και οι υπόλοιπες 11 με 13 συμφωνίες είχαν διάφορους περιορισμούς. Πού μπορούσαν να πάνε οι, να, οι κλπ. Η καναδική πολιτική έγινε όλο και πιο φιλελεύθερη σταδιακά τώρα ε, ακολουθεί μια πολιτική των γαλαζίων, γαλάζιων ουρανών. Πριν όμω ήταν πολύ περιοριστική και κάποιε από τι καναδικέ συμφωνίε εξακολουθούν να παραμένουν. Παραδείγματο χάρη, ο Καναδά είχε πολύ αυστηρέ πολιτικέ, περιόριζε τα, πέμπτα, τα δικαιώματα του πέμπτου τομέα ε, σε διάφορα σημεία της Αμερική. Υπό αυτές τις περιστάσει, η προστιθέμενη αξία μια συμφωνία Καναδά και Ευρωπαϊκή Ενώσεως ήταν πολύ μεγάλη και η συμφωνία του 2009 οδήγησε στα αποτελέσματα όσον αφορά τα δικαιώματα κυκλοφορίας. Θα σημειώσω το ότι οι τελευταίες δύο κατηγορίες, μόνο οι δύο τελευταίες κατηγορίες, δεν παρήγαγαν κάποια αποτελέσματα. Οι άμεσες υπηρεσίες που πριν ε, περιοριζόταν πάρα πολύ αυστηρά, στις περισσότερες διμερείς συμφωνίες, τώρα έχουν απελευθερωθεί πλήρως Όμω, όπω αναφέρω και στο ενημερωτικό μου σημείωμα η, η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά δεν προχωρεί τόσο μακριά όσο η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση είπα όσον αφορά τα δικαιώματα κυκλοφορία και πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά. Γι' αυτό η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά α, προβλέπει σταδιακή εισαγωγή των μέτρων και εδώ έχω ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποθέσεις που ακολουθεί το κείμενο, αντικατοπτρίζονται στα παραρτήματα της εν λόγω ο Καναδά έχει κίνητρα να χαλαρώσει του ελέγχου όσον αφορά τι ξένε επενδύσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αντάλλαγμα, με νέα δικαιώματα πέμπτη κατηγορία του Καναδά στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, απεριόριστα δικαιώματα που, που απολαμβάνει ο Καναδά ε, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέραν αυτών. Λοιπόν, είναι πολύτιμα, περισσότερο πολύτιμα τα δικαιώματα τη πέμπτη κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι για του Καναδού. Λοιπόν, συγκρίνοντα τι δύο συμφωνίε, δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα δεν έχουν κίνητρα είπα, ούτε ο καναδα να προχωρήσουν στι παραπέρα φασει τώρα στην οικονομική συγκυρία. Τώρα ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Πώ μπορεί να ενεργοποιηθεί ο διάλογο στον αφορά αερομεταφορέ. Μια πιθανότητα είναι στι συζητήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώση είπα, ή στην, να μπει το θέμα τη βορειοατλαντική απελευθέρωση αγορά. Αυτό ο διάλογο πρέπει να εστιάζεται περί συνεργειακών ε, ποιοτικών ελέγχων και να υπάρχει ευαισθητοποίηση. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι είναι δημόσια αγαθό η αερομεταφορά και χρειάζεται και εξαρτάται η αποδοτικότητα του εμπορίου και του ταξιδίου σε αυτό το τομέα, κυρίως όσον αφορά τις επενδύσεις. Είναι βασικό στόχο θα μπορούσε να είναι εξή. Ε, να διαπραγματευτούμε έναν τρόπο για κλασικέ εξαιρέσει στο τομέα των μεταφορών και να πολεμήσουμε για εθνική αντιμετώπιση των θεμάτων όσον αφορά τι επενδυτέ των αερομεταφορών, όπω γίνεται για όλου του άλλου τομεί τη οικονομία. Νομίζω ότι θα έχουμε ρωτήσει αργότερα, οπότε θα κάνω μία τελική παρατήρηση. Ένα ερώτημα που έθεσε η διαπραγματευτική, δημιούργησε η διαπραγματευτική διαργασία με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά αφορούν διαπραγματεύσει την ίδια χρονική περίοδο και την ίδια περιοχή. Αλλά θεωρούνται σαν δύο ανεξάρτητε, τελικά εκτελήφθηκαν σαν δύο ανεξάρτητε διμερεί διαπραγματεύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε παρόμοια προσέγγιση. Υπάρχουν όμω διαφορέ φορολογικέ και διαθωτικέ. Ε, και αυτό φαίνεται στι συμφωνίε. Και ίσω κάτι που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατυπώνει τι εντολέ τη επί τη βάση ε, προτύπων στόχων που μπορεί να αντικατοπτρίζονται σε ένα πρότυπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τι συμφωνίε, ή θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένε περιπτώσει κάθε φορά εντολή που δίνει σε διαπραγματεύσει. Λοιπόν, ε, μπορώ να ακούσω ερωτήσει τώρα ή μετά αφού κάνει παρουσίαση και δύο συνάδελφοι. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στάινεν. Θα ακούσουμε πρώτα τους καλεσμένους μας και μετά θα γίνουν ερωτήσεις. Αλλά σας ευχαριστώ που εμείνατε στο χρόνο σας. Ο κύριος Κλότ Πρόπστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με προσκάλεσε για την παρουσίαση αυτή. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μια αξιολόγηση, όπως μου ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της προστιθέμενης αξίας ε, των ε, συμφωνιών που συνήψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει κάτι τέτοιο, για να γίνει αυτή η αξιολόγηση, αναζήτησα κάποια κριτήρια και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη της ανακοίνωση το 2002, μετά την απόφαση του ΔΕΚ, είναι να προσδιορίσει ίδια κάποιους στόχους Βλέπετε τους στόχους σας στην διαφάνεια, δεν πρόκειται να τις μεταφράσω τώρα από τα αγγλικά στα γαλλικά. Και μια και οι στόχοι αυτοί έμειναν αμετάβλητοι στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι καλό σημείο αναφορά για να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι συμφωνίες ε, υλοποιούσαν αυτούς τους στόχους και άρα παρήχαν την αναμενόμενη προσθεθέμενη αξία. Αν εξετάσουμε τον πρώτο στόχο, ήταν ε, νομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, οι συμφωνίες που συνήθισαν επιτρέπουν την προσαρμογή των διμερών συμφωνιών που είχαν συναυθεί από τα κράτη-μέλη προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με το κοινοτικό δίκαιο. Η απάντηση είναι καταφατική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθισε 55 οριζόντια συμφωνίες με τρίτες χώρες, συμφωνίες που ε, τροποποιούν αμέσως όλες τις προϋπάρχουσες συμφωνίες και τις ευθυγραμμίζουν με το κοινοτικό δίκαιο. Οπότε είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο και λειτουργεί πολύ εύρυθμα. Το σύνδεσμο πρόβλημα στην αεροπορία είναι ότι οι διμερείς συμφωνίες γίνονται μόνο μεταξύ ε, συμβαλωμένων μερών που το επιθυμούν. Δεν γίνεται διαπραγμάτευση με χώρες που δεν θέλουν να συνάψουν συμφωνία. Ε, με χώρες που δεν θέλουν τη ρήτρα για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τους πείσουμε λοιπόν διμερώς. Μπορούμε να βρούμε κάποια μέσα πίεσης, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματικά αυτά. Οπότε το διμερές σύστημα έχει κάποια όρια. Ένα άλλο μικρό πρόβλημα είναι ότι μερικές χώρες θεωρούν ότι για να γίνει μια κοινοτική αεροπορική εταιρεία, για να δικαιούται δικαίωμα μεταφορά τη διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρε θα πρέπει να έχει έδρα στο έδαφος αυτή της χώρας και δεν ξέρουμε αν αυτό είναι συμβατό με την οδηγία για τι υπηρεσίε. Οπότε οι οριζόντιες συμφωνίες επιτρέπουν την ευθυγράμμιση των διμερών συμφωνιών των κρατών μελών με το κοινοτικό δίκαιο αλλά ίσως εξαιτία της πρακτικής ε, τρίτων χωρών δεν αξιοποιούν στο έπακρο το δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο στόχο. Ο δεύτερος στόχος, όπως ε, το διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνίσταται σε μια πολιτική μεταρρύθμιση του διεθνού συστήματος προκειμένου να προωθηθούν οι αεροπορικές ε, υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων ώστε να γίνουν επενδύσει στον τομέα των αερομεταφορών. Ο στόχο αυτός παρτίζεται από δύο σκέλη. Καταρχήν θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν οι συμφωνίες όντως συμβάλλουν στην πρόθεση των αερομεταφορών και θα ξεκινήσω από αυτό το, το σκέλος. Γιατί μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι δύσκολο να αποδείξουμε με αδιάστατα επιχειρήματα το κατά πόσο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές εταιρείες συνέβαλαν στην πρόθεση των αερομεταφορών. Αναζήτησα κάποια στατιστικά στοιχεία και μόνο από τη Eurostat τα βρήκα κάποια στοιχεία. Και στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε και που κυκλοφόρησε από τη γραμματεία του Κοινοβουλίου βλέπετε διάφορες καμπύλες που προσπαθούν να συγκρίνουν την κατάσταση μεταξύ των χωρών που έχουν παρόμοιες αγορές για να δούμε αν οι αερομεταφορές ε, αναπτύχθηκαν γρηγορότερα με τους κυρωτικούς εταίρους ή με τους υπόλοιπους. Η απάντηση είναι αρνητική. Δεν μπορούμε σήμερα να ισχυριστούμε ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες συνέβαλαν πραγματικά στην προώθηση ε, και στην σημαντική ανάπτυξη των αερομεταφορών, με μία εξαίρεση, το Μαρόκο διαπιστώνουμε ότι η εξέλιξη των αερομεταφορών στο Μαρόκο προηγείται τη σύναψη συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον οφείλεται στην ε, πολιτική της μαροκινής κυβέρνησης για απόλυτη απελευθέρωση των ε, αεροπορικών μεταφορών. Δεν ήταν λοιπόν ε, αποτέλεσμα της συμφωνίας με, το, με την κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις, τα, τους ναύλους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια μελέτη που εκπώνησε, την οποία δεν είδα, λένε ότι ε, συνέβαλαν όντως ε, οι δομές των ε, ναύλων, αλλά είναι περίπλοκες αυτές οι δομές για να συνάψουμε κάποια συμπεράσματα και θα πρέπει και πάλι να κάνουμε σύγκριση με την κατάσταση χωρών που δεν έχουν τέτοιες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση και μας ε, το επισήμανε και ε, ο κύριος Φωνστάιν για τις συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και τον Καραδά. Το θέμα είναι οι συμφωνίες αυτές ε, προβλέπουν νέα δικαιώματα, αλλά αξιοποιούνται, ασκούνται αυτά τα δικαιώματα. Ή... Δημιουργήθηκαν νέοι προορισμοί, νέες μεταφορές. Τα στοιχεία της Eurostat δεν μας βεβαιώνουν για κάτι τέτοιο. Και η εξέλιξη των υπηρεσιών ε, χωρών που έχουν συμφωνίες δεν ήταν διαφορετικές από ε, ε, την εξέλιξη υπηρεσιών ε, προς χώρες που δεν έχουν συμφωνίες. Τώρα, αυξήθηκαν οι επενδύσεις χάρη στις συμφωνίες ή διευκολύθηκε η διακίνηση των κεφαλαίων. Ο κύριος Φωνστάινεν απάντησε αρνητικά σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Βέβαια, ο Καναδάς έχει διαφορετικό σύστημα που προβλέπει ότι μπορούμε να έχουμε αμοιβέ επενδύσει στις αεροπορικές εταιρείες υπό την επιφύλαξη όμως ότι ο Καναδάς θα τροποποιήσει την νομοθεσία, κάτι που τελικά δεν έκανε. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες συμφωνίες που συνήθισαν με τη Γεωργία, την Ιορδανία, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερο μηχανισμό για αμοιβέ επενδύσει στις αεροπορικές εταιρείες. Απλώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ανακύψει το θέμα θα εξεταστεί περιπτωσιολογικά και έχουμε και μικτές επιτροπές που προβλέπουν οι συμφωνίες. Η μόνη συγκεκριμένη περίπτωση όπου διαπιστώθηκε άνοιγμα προς την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι η συμφωνία που έγινε ε, ΕΚΑ που αφορά ενιαίο πυλώνα που είναι παρόμοια με τη συμφωνία που έγινε με την Ελβετία και που δίνει παρόμοια αποτελέσματα με τη συμφωνία των δύο πυλώνων που συνήψαμε με την Ισλανδία και την Ορβηγία. Εκεί έχουμε ένα είδος προένταξης, χωρών δηλαδή που κάποια στιγμή θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδέχονται το σύνολο του κοινοτικού δικαίου και την ομολογία του ΔΕΚ και τις εξουσίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας. Οπότε ούτε για τις επενδύσεις έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρίτο στόχο, την ε, πρόθεση του ανταγωνισμού. Όλες οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπουν επιπλέον ε, δικαιώματα με διατάξεις και μηχανισμούς για τους ναύλους, για τις τιμές, για το δυναμικό που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το θέμα είναι όμως ότι αυτές οι συμφωνίες συνήθισαν με φιλελεύθερους εταίρους που παρήχαν αντίστοιχα δικαιώματα μέσω των διμερών συμφωνιών. Οπότε αν θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό θα πρέπει ε, να διαπραγματευτούμε με χώρες που είναι πολύ λιγότερο φιλελεύθερες και για τις οποίες ε, θα έχει κάποιο στόχο η ο κοινοτικό κλάδος, ο ευρωπαϊκός κλάδος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις λοιπές διατάξεις που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού, θα ήθελα να πω ότι πέραν τη συμφωνίας με τις χώρες των Βαλκανίων, που θέλουν να εξομοιωθούν με τις ευρωπαϊκές χώρες και άρα δέχονται το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου για θέματα ανταγωνισμού και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπόλοιπε συμφωνίε ελάχιστε διατάξει ε, περιλαμβάνουν προ την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν κάποιε διατάξει για τι κρατικέ ενισχύσει που συνήθω λένε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό για τον ανταγωνισμό και αν υπάρχει πρόβλημα θα συνεργαστούμε να το λύσουμε. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη ή μηχανισμό που να προβλέπει εκ των προτέρων να προβλέψουμε τι θα συμβεί σε περίπτωση αντιδικία, αντιπαράθεση. Οπότε ούτε και εδώ είμαι βέβαιος ότι οι συμφωνίε συμβάλλουν στην πρόθεση του ανταγωνισμού στις αερομεταφορές. Τώρα, σε ό,τι φορά τον τέταρτο στόχο, που αφορά την κανονιστική σύγκληση. Προσπαθήσαμε να πείσουμε ε, κάποιες χώρες να ευθυγραμμίσουν την νομοθεσία τους ε, με την ε, κοινοτική και να ρυθμίσουν και τις ε, αεροπορικές μεταφορές και ροές. Ε, διατάξεις για την ασφάλεια, την προστασία. Είναι κάποιες στερεότυπες διατάξεις που σταθερά περιλαμβάνονται στις διμερείς ε, συμφωνίες και δεν προσθέτουν και τίποτα. Ούτως ή άλλως οι χώρες αυτές δεν θέλουν να ευθυγραμμίσουν την ομοθεσία τους με την κοινοτική. Εδώ και δεκαετίες έχουμε συζητήσεις με τους Καναδούς, τους Αμερικανούς, τους Βραζιλιάνους για την εναρμόνιση, τη σύγκληση, την κανονιστική, αλλά είναι μια διαδικασία που είναι τελείως ξεχωριστή από τη σύναψη των συμφωνιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λοιπές συμφωνίες, τις συμφωνίες που συνάπτουμε με γειτονικέ χώρες, εκεί υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις που προβλέπουν ευθυγράμμιση της ε, νομοθεσίας τους με την κοινοτική κάποιες μεταβατικές διατάξεις που συνδέουν την χορήγηση των επιπλέον δικαιωμάτων της, της πέμπτης ελευθερίας ή του καμποτά στην κοινότητα με την πρόοδο που έχει συνηθίσει σε θέματα ευθυγράμμισης της νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο, της κανονιστικής σύγκλησης δηλαδή. Η διαδικασία αυτή μεταβατική είναι αρκετά περίπλοκη και για να αποκτήσει κανεί τα επιπλέον δικαιώματα, θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει ότι όντω η χώρα αυτή ευθυγραμμίστηκε με το κοινοτικό δίκαιο, ότι έχει επέλθει αυτή η κανονιστική συγκλήση και η διαδικασία αυτή είναι υπερβολικά χρονοβόρα. Και μια και τα δικαιώματα των μεταφορών ε, δεν έχουν και πολύ σημαντική οικονομική αξία, δεν είναι και επιχείρημα ε, υπέρ της κανονιστικής σύγκλησης. Η μόναδική περίπτωση όπου είχαμε πραγματική ε, σύγκληση και δυνατότητα με τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά οι περισσότερες χώρες ούτως ή άλλως συμμετείχαν στη Eurocontrol, στην, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον έλεγχο της αεροπορίας και ούτω καθεξής. Οπότε ήδη οι χώρες αυτές είχαν ξεκινήσει την ευθυγράμμιση. Επίσης ζητάμε από τις χώρες να ευθυγραμμιστούμε το κοινοτικό δίκαιο, αλλά δεν τους λέμε με ποιο τρόπο να το κάνουν. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία, ήμουν διευθυντής της ΆΖΑ για κάποιο χρόνο και ζητάμε από τις, χώρες, τις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία ε, για θέματα ασφάλειας αλλά τους επιβάλλουμε και τα δικαιώματα της Επιτροπής ή της ΆΣΑ. Αλλά καμία χώρα δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι η ΆΣΑ θα πρέπει να ε, εκδώσει πιστοποιητικό ασφάλεια για τα αεροπλάνα του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι τι διαιτητής σε περίπτωση αντιπαράθεσης ή αυτέ φιλονικίες. Οπότε έχουμε χώρε κατάλογο κανονισμών που θέλουμε να τηρήσουν τρίτες χώρες, αλλά ο σε περιπτωση αντιπαράθεση κάποιε φιλονικιε οποτε εχουμε ενα καταλογο κανονισμων που θελουμε να τηρησουν οι τριτες χώρε, αλλα ο στόχο αυτό δεν είναι και πολύ σαφής, γιατί στον κατάλογο περιλαμβάνονται και κανονισμοί που οι τρίτες χώρες δεν θέλουν να εφαρμόσουν. Τώρα για τα συμπεράσματά μου. Θα ήθελα να σας πω εν συντομία ότι είναι σαφές ότι οι οριζόντιες συμφωνίες έχουν ε, μια προστιθέμενη αξία για να, και για να διευκολύνουν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν ε, περιορισμούς ή δεν επιβάλλουν την υποχρεώση έδρας ε, στο έδαφος τους για να τη θεωρήσουν κοινοτικούς οι συμφωνίε με τα Βαλκάνια είναι καλέ, αλλά οι μεταβατικοί μηχανισμοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι και σε ορισμένε περιπτώσει αναχαιτίζουν την πρόοδο σε ό,τι αφορά την κανονιστική σύγκληση σε ορισμένου τομεί. Στον τομέα τη ασφάλεια τη αεροπορία, για παράδειγμα. Κάποιε χώρε θα μπορούσαν να είχαν εξομοιωθεί με τι κοινοτικέ χώρε των Βαλκανίων, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν έχει τεθεί σε ισχύ ακόμη συμφωνία. Του ζητούμε να περιμένουν τις κανονιστικές συγκλήσεις και σε άλλους τομείς. Οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες αυτές ε, λίγα πράγματα προσφέρουν σε σχέση με τις υπάρχουσες ε, διμερείς συμφωνίες. Και για να δούμε κάποια πρόοδο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση να διαπραγματευτεί με λιγότερο φιλελεύθερες χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι αν έχουμε διαπραγματεύσει με τις λιγότερο φιλελεύθερες χώρες θα επιβληθούν περιορισμοί σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, το δυναμικό τα σημεία εξυπηρέτηση και το πόσο, πώς θα γίνει η κατανομή των δικαιωμάτων μεταξύ των αερομεταφορέων, ούτε και αυτό είναι προφανές πώς θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι χώρες αυτές ε, δεν έχουν καν πρόθεση να διαπραγματευτούν τέτοιε συμφωνίες με την ε, κοινότητα. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν οι στόχοι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούνται. Αν δεν υλοποιούνται θα πρέπει να βρούμε άλλο σύστημα πλέον του διμέρους ίσως τα θέματα των αεραμεταφορών να τα διαπραγματευτούμε ταυτόχρονα με άλλα ζητήματα, είτε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, είτε στα πλαίσια διμερών συμφωνιών πολυτομεακών, πολυκλαδικών, ώστε ε, ό,τι χάνεται σε ένα τομέα να ανακτάται σε άλλο και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείστε και το μικρόφωνο. Ευχαριστώ ο κύριος Ατά Χουσέιν Χάν, κατόπιν Γενικός Γραμματέας ε, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ πέρα για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις απόψεις της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών για την ε, συνολική πολιτική εξωτερικών αεροπορικών μεταφορών και έχουμε δώσει τίτλο εδώ πέρα ε, στην πολιτική αυτή το να ξαναβάλουμε την Ευρώπη στον χάρτη. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές ε, προσθέτουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία την ημέρα. Την ημέρα. Απασχολούν 5 ε, εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και αν α, ε, λάβουμε και τη δεύτερη περιφέρεια, δηλαδή του Ευρωπαϊκού και άλλες εταιρείε, ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 8 με 9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρουν γύρω στα 800 εκατομμύρια επιβάτες το έτος και στην Ευρώπη και διεπιρωτικά. Οπότε είναι σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τώρα, εξακολουθούμε να θεωρούμε, και το βλέπετε εδώ πέρα, πως ε, ο διαχειριστής ε, του δικτύου και οι μεταφορές μέσω μεγάλων κόμβων είναι ο βασικός τρόπος μεταφοράς ε, επιβατών και αγαθών ε, ανά την Φίλιο. Αν δείτε εκεί πέρα στη μέση βλέπετε πως υπάρχει ένα επίπεδο πολλαπλασιαστή και ο τρόπος ο οικονομικά αποτελεσματικός είναι με κόμβους ε, που θα έχουν διπυρωτικές συνδέσεις. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε πως, να συνειδητοποιήσουμε πως 30 με 35% των Ευρωπαίων επιβατών κάνουν πτήσεις με πολλά σκέλη για να πάνε στον προορισμό τους και τέλος οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προωθούν και έχουν α, τέσσερις φορές περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις μη ευρωπαϊκές εταιρείες. Ένα μεγάλο λοιπόν επιχείρημα για το να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Τώρα θα σας ε, πω πώς βλέπουν την αεροπορία σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί όπως σας είπα χρειαζόμαστε μεγάλα αεροδρόμια για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε πως γίνονται επενδύσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, κυρίως Μέση Ανατολή και από Ανατολή και σας διαβεβαιώ πως τα στοιχεία με την ε, Ινδική υποήπειρο και την Νότια Αμερική τα ίδια νούμερα θα δώσουν. Δυστυχώς η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτές τις επενδύσεις και αυτό μας ανησυχεί αν θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε ε, αυτή την διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Να μπούμε τώρα λίγο σε λεπτομέρειες. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια τέτοια συνολική πολιτική αρματοφόρων. Πρέπει πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Δεν έχει νόημα να διαπραγματευόμαστε διεθνώς διεθνείς συμφωνίες όπως ανέφεραν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές χωρίς να έχουμε κάνει τα βασικά στην Ευρώπη οι ε, ευρωπαϊκές αναμεταφορές ε, εξακολουθούν να είναι οι πιο βαριά φορολογούμενες ε, στον κόσμο και οι πιο πολύ ρυθμιζόμενες και δεν είναι σωστό αυτό για την ανταγωνιστικότητά τους. Έχουμε λοιπόν κάποιους, ανταγωνισμούς, κάποιους κανονισμούς που αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις και ε, τη ξεκίνημα νέων εταιριών που δεν εφαρμόζονται δυστυχώ ε, πάντα. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν είναι αποτελεσματικέ υποδομέ. Αναφέρθηκα σε υποδομέ στο έδαφο, αλλά ε, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός αφορά και υποδομές στον ουρανό. Και τέλο πρέπει να δούμε τα παγκόσμια ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και βασικό παράδειγμα προφανώ είναι να ε, δούμε την συμπερίληψη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών, το οποίο πλέον ευτυχώ θα αντιμετωπιστεί στο επίπεδο του ΙΚΑΟ. δούμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει στο ε, επίπεδο το διεπηρετικό. Πρέπει να βασιστούμε σε ξεκάθαρα επιχειρηματικά μοντέλα. Μόλις ανέφερε ο συνάδελφο το ότι πολλές από τι ημερείς συμφωνίε ε, δεν έχουν προχωρήσει τόσο όσο αρχικά ελπίζαμε και κάποιε δεν είχαν το όφελο που θα θέλαμε. Οπότε πρέπει να είμαστε σαφείς και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κάνουμε αξιολόγηση. βεβαίω, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, το είπα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως δεν ε, έχουμε συμφωνία αερομεταφορών ε, η οποία θα είναι για κάθε ε, εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, δημιουργικοί στο να προσαρμοζόμαστε ε, στις ιδιαιτερότητες της κάθε τρίτης αγοράς. Δεν υπάρχει μία λύση μόνο και οπωσδήποτε όχι στην τρέχουσα κατάσταση. Υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια λοιπόν που θα θέλαμε να, να σας αναφέρουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού στο διεθνές επίπεδο. Όπως είπα, να γίνει μια σαφής ανάλυση χωρίς προκαταλήψεις. Όπω ε, ε, όπως είπα προηγούμενος ο μιλητής, ανέφερε κάποια πράγματα, να εστιάσουμε σε μια σύγκληση και εναρμονισμό των κανόνων. Σημαντικό αυτό για ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αντιλαμβάνω βεβαίως, αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω πως όσον αφορά το περιβάλλον, τα δικαιώματα των επιβατών και ίσως και την ασφάλεια υπάρχουν κάποιοι τομεί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, όπως είπα, δεν υπάρχει μία ενιαία λύση. Πρέπει λοιπόν να δούμε και νέους τύπους συμφωνιών με τρίτες χώρες όταν δεν υπάρχει προφανώς αμοιβαίο όφελος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο διμερές περιφερειακό και στο επίπεδο του ΙΚΑΟ. Τέλος, πρέπει να, είναι, ε, να είμαστε σαφείς στην απελευθέρωση της ιδιοκτησίας και ελέγχου. Εάν δείτε την ε, συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε πως οι Ευρωπαϊκέ εταιρείε επιτρέπουν 49% ξένη ιδιοκτησία ενώ στην Αμερική επιτρέπεται μόνο 25% ξένη ιδιοκτησία. Πρέπει να είναι σαφές πως ε, αυτά τα πράγματα ε, θα είναι κρίσιμα στο προσεχισμένο. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι ο θεμητό και δίκαιος ανταγωνισμός. Αυτή, στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πως ε, βλέπουμε εμείς τον θεμητό ανταγωνισμό. Εποπτεία του ανταγωνισμού, ανεξάρτητες αρχές, έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων, διαφάνεια των λογαριασμών και όσον αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο διαφόρων παρόχων, να, σχετίζονται, να σχετίζονται το κόστος με την παροχή των υποδομών και προφανώς μη διάκριση στην πρόσβαση των υπηρεσιών για όλους σε αεροδρόμια εκτό Ένωση. Αυτά έτσι ω κάποιες πρώτες παρατηρήσεις και οπωσδήποτε αναμένω τις ε, ερωτήσεις σας και την συζήτηση με τον εισηγητή, τον κύριο Μαρινέσκου, για την ε, εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καν. Λοιπόν, όποιος θέλει να αποβάλει ερώτηση, σηκώ στο χέρι του. Ο κύριος Κούν για το ΕΛ ξεκινά. Θα ακολουθήσω τη σειρά των ομάδων. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές. Κύριος και Πρόστ. Ήταν ενδιαφέρον ε, να δούμε το βαθμό της πολυπλοκότητας που υπάρχει εδώ πέρα. Εγώ αντιλήφθηκα πως υπάρχουν πάρα πολλά σημεία αναφέρα τις εμπορικέ συμφωνίες με ΙΠΑ και Καναδά, αλλά και την ασφάλεια πτήσεων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίως Ευρωπαϊκός Ουρανός, αλλά και εκεί όπου προσπαθούμε, αλλά δεν γίνεται ε, κάποια πρόοδος, δηλαδή στα airspace blocks, την ασφάλεια, το εάν έχουμε την απαγόρευση ή αλλά πράγματα ειδικά όταν μιλάμε για διπυρωτικέ πτήσει, ο κύριος Χάν σωστά είπε πω πρέπει να δημιουργηθεί κάποια τάξη, να υπάρξει μια τάξη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και στο εσωτερικό και σε κάποια κράτη-μέλη είμαστε λίγο πίσω. Εδώ λοιπόν Μιλήσατε για ένα δισεκατομμύριο ευρώ την μέρα, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ευκαιρίες δηλαδή για ανάπτυξη που δεν επιτρέπεται να χάσουμε στην Ευρώπη. Ειδικά δεδομένη οικονομικής κατάστασης. Μεταφορά αγαθών και επιβατών μεταξύ των μεγάλων εμπορικών κόμβων ε, Βορειοαμερική, ΗΠΑ, Καναδά και ε, Νότιο-Ανατολική Ασία μέσω Ντουμπάι ε, αυξάνεται, το είπατε, και πρέπει και εμείς να ε, λάβουμε μέρος. Και το θέμα του εμπορίου και των ζωνών ελευθερου μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρθηκε. Το τι, τι επιπτώσεις θα έχει στο δικό μας το θέμα είναι σημαντικό. Εμπορία εκπομπών. Και εδώ πέρα ένα σημείο τριβής. Έχουμε κάποια πιθανότητα δεδομένης της πτώσης της τιμής ε, του διοξιδίου του άνθρακα να επιτύχουμε στόχους που πρέπει βέβαια όλα αυτά να τα δούμε σε σχέση με τον δίκαιο ανταγωνισμό και τι ρόλο παίζει και ο ΠΟΕ στις διαπραγματεύσεις κάνουμε διμερός για το θέμα αυτό. Για τις υποδομές το αναφέραμε για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και τους μεγάλους κόμβους και το ότι παίζουν ένα μεγαλύτερο ρόλο δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά. Επενδύσεις στις υποδομές, το εάν μιλάμε για σιδηρόδρομους, ε, οδικές μεταφορές ή ε, αεροδρόμοι ε, αποτελούν πάντα προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Και το σημειώνω αυτό που είπατε. Και εδώ πέρα έχει, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε από κοινό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλεχαντραουή Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές για την εισαγωγή τους που δεν είναι έτσι τόσο θετική αλλά τα συμπεράσματα είναι πως οι προσδοκίες ε, δεν ε, υλοποιούνται. Εγώ δεν πίστευα τόσο πολύ στα δισεκατομμύρια κερδών που προέβλεπε η Κομισιόν στην ανάλυση της. Η κρίση, ε, νομίζω η γενική οικονομική κρίση, μήπως δυσκολεύει το να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τώρα ήδη. Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας. Δεύτερον, όσον αφορά την σύγκληση των κανόνων. Σημαντικό αυτό. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε, π.χ οι μεγάλες διαφορές ε, στις συνθήκες εργασίας, στους μισθούς, σε ένα τομέα που θα έπρεπε να είναι λίγο πολύ ίδιοι. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για αριθμιστική σύγκληση, μιλάμε για τρίτες χώρες. Τι, πώς το βλέπετε συγκεκριμένα, ποια είναι τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία, στα οποία θα πρέπει να συγκλίνουμε. Και μετά από αυτό, για να φύγουμε από τις συζητήσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοιων χωρών. Δεν υπάρχει κάποιος ε, ρόλος και για τις αεροπορικές εταιρείες μέσω των συμμαχιών τους για να γίνουν συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο σε κάποια πράγματα εντός μιας αεροπορικής συμμαχίας. Παραδείγματο χάρη γίνονται συνομιλίες στο πλαίσιο του ETS, παραδείγματο χάρη, μεταξύ αεροπορικών εταιριών για να δημιουργηθεί μια, να διαμορφωθεί μια κοινή θέση. Ε, αυτό ισχύει και για κάποια άλλα θέματα. Τέλος, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, Θα ήθελα να δω συγκεκριμένα την σύγκριση μεταξύ αυτού που γίνεται παραδείγματο χάρη σε ένα αεροδρόμιο στη Μέση Ανατολή και των εταιριών αυτής της περιοχής και της δικής μας προσέγγισης στην Ευρώπη, ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Α, υπάρχει κάποια απογοήτευση γιατί όλο ακούμε πως υπάρχουν δισεκατομμύρια κερδών που θα επιτύχουμε και δεν τα βλέπουμε πουθενά. Αλλά σε αυτό στο οποίο συμφωνείτε είναι πως με τις νέες ε, συμφωνίες δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το πλεονέκτημα ότι έχουμε κάποιες συμφωνίες γιατί με κάποια κράτη δεν είχαμε καθόλου. Οπότε θα έχουμε την ίδια, αν και όχι ίσως ε, πάρα πολύ καλή κατάσταση συγκεκριμένα, για την συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εδώ πέρα ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλήξουμε σε μια τέτοια ισότιμη σχέση γιατί οι ΙΠΑ πάντα έχουν πλέον εκτήματα. Ο κύριος Χάν αναφέρθηκε σε... στο ζήτημα της ιδιοκτησίας όπου επιτρέπεται ξένη ιδιοκτησία στις ΙΠΑ να είναι 25% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 49%. Εγώ ήμουν τότε όταν είχαν πάει στην Ουάσιγκτον νέα και αισιόδοξη βουλευτής ε, και τους είχα πει πως θα κάνουμε και εμείς κάποιες παραχωρήσεις αν ανεβάστηκε σε αυτό το ποστό. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει ποτέ ισότητα γιατί όταν θέλουμε εμείς κάτι τε ζητάνε κάτι παραπάνω συνέχεια είπα. Θα παραμείνει λοιπόν αυτή η διαφορά. Γι' αυτό είχαμε σκεφτεί το εάν πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ανισορροπία ταυτόχρονα. Βέβαια, είναι μεγάλος εταίρος είπαμε τεράστιο ποσοστό των παγκοσμίων αερομεταφορών. Οπότε το ζήτημα τώρα είναι, θεωρείτε πως θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Ίσως αν οδηγηθούμε σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Ομπάμα σε μια ομιλία του. Και όσον αφορά τον Καναδά, έχω την εντύπωση μετά την παρουσίαση του κυρίου Φονταστάινεν πως υπάρχουν κάποια πλέον εκτήματα. Το τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Χάν. Μιλήσατε για ίσους ανταγωνισμού και είπατε πως πρέπει να σκεφτούμε νέους τρόπους συμφωνιών με τρίτες χώρες αν δεν υπάρχει αμοιβαίο οικονομικό όφελος. Πώς α, το βλέπετε και αυτό θα μπορούσε να είναι και μια υπόδειξη ίσως προς την Κομισιόν. Τι βελτιώσει θα μπορούσαμε να επιφέρουμε. Αυτά και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε και εμείς θα θέλαμε να μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπέργκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο τις ε, φοβερές ε, υποσχέσεις για τα οικονομικά ωφέλη των συμφωνιών αυτών που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν να ε, τσεκάρουμε, να δούμε τι γίνεται και τι μας είχε υποσχεθεί τότε η Κομισιόν ως οικονομικό αποτέλεσμα. Δεύτερον, συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Θεωρώ πως σε ένα συγκεκριμένο τομέα είναι προβληματική. Στην τελευταία μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Ελχαντραούι νομίζω είχαμε συζητήσει επί μακρόν για το εάν έχει νόημα εφόσον η ΕΠΑ συνεχώς ε, έχουν νέες απαιτήσει για να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, αν έχει νόημα να διαπραγματευόμαστε. Αυτό το οποίο παρατηρώ εγώ είναι πως εδώ πέρα δεν υπάρχει ετοιμότητα να υπάρξουν ε, ίσοι όρια Είναι προφανές. Και πρέπει να σκεφτούμε το τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία. Ξέρω βεβαίως πως ε, συζητάμε μόνο τις, ε, τις κρίσιμες ε, περιπτώσεις, αλλά σκέφτομαι το τι θα γίνει παραπέρα. Όταν συζητάμε για ρυθμιστική σύγκληση παγκοσμίως, και μιλάμε για μισθούς ασφάλεια ή το οτιδήποτε. Αν δούμε κάποιες περιοχές του κόσμου και μετά έχουμε την ελπίδα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια, τους μισθούς ε, και τις συνθήκες εργασίας και το χρόνο πτήσης θεωρεί πως ε, μπορεί να να κάνει ό,τι θέλει τις υπόλοιπες ε, μεγάλες ε, δυνάμεις στον, στον τομέα αυτόν. Δεν ξέρω πως θα νερωθεί τελικά τα, οποία, αυτά τα οποία έχουμε και ισχύουν εδώ πέρα στην Ευρώπη. Και όλα αυτά υπό τον τίτλο «Ναι, εντάξει, μπορεί να βγάλουμε κανένα φράγκο». Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που μου ασχολούν εμάς στον τομέα της αεροπορίας ε, δεν λαμβάνονται υπόψη. Παριστάνουμε συνεχώς πως υπάρχουν μόνο θετικά αποτελέσματα. darf, was die Kollegin Meissner gesagt hat in Bezug auf die ähm, Forderung, die Nachtflugbeschränkungen für και μας ζητάτε να μειωθούν οι περιορισμοί στις αεροπορικέ εταιρείε των ΗΠΑ για να γίνει κάτι παραπάνω. Μονίμω για να γίνει κάτι παραπάνω. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το θέμα στο μέλλον και εδώ πέρα η Κομισιόν πρέπει να το δει το πράγμα. Όχι μονίμως να έχει τα μάτια της γεμάτα δολάρια. Κυρία Φώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους φιλοξενούμενους μας για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Πριν προβώ σε σχόλια. Έχουμε αυτό το βιβλιαράκι εδώ, αυτό το φυλάδιο. Αναφέρει τις συμφωνίες για τις ε, υπηρεσίες ε, αεροπλοείας. Δεν υπάρχει πλήρης κατάλογος ε, των συμφωνιών Αναφέρθηκαν κάποιες, δεν αναφέρονται εδώ λεπτομερώς, αναφέρθηκαν κάποιοι τομείς και κάποιες περιοχές. Πριν από καιρό το είχαμε κουβεντιάσει αυτό, Πρόεδρε, θα το θυμόσαστε. Μα είχαν πει ότι θα είναι η πανάκια. Από διμερεί έπρεπε να προχωρήσουμε στα εκεί. Ε, δεν διαφωνώ. Πρέπει να δει κανεί τι πρακτικέ πτυχέ. Δεν θεωρούσα ότι θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Θα αναφερθώ σύπα αργότερα. Διότι όλα εκεί εστιάζονται. Εγώ θα έλεγα μην σαστούμε παρά αποκλειστικά εκεί, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τη Βραζιλία. Μεγάλη αγορά είπα, αλλά είπα κάνα και συμφωνία με τη Βραζιλία. Εμεί όχι. Με την Κίνα τι γίνεται. Ρωσία, Ινδία, τεράστιε αναδυόμενε αγορέ. Σημαντικότατε θα είναι. Ενημερώστε μα παρακαλώ. Βέβαια, λαμβάνοντα υπόψη το τι μπορείτε να αναφέρετε δημοσία. Αναφέρθηκα κάποιες συμφωνίες, θα ήθελα λεπτομέρειες. Έχουμε το έντυπο, όπως προανέφερα. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΙΠΑ. Έχουμε ξεκινήσει από παλιά αυτή την προσπάθεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα πάρουν περισσότερα ακόμα. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Οι καλοί μας φίλοι στη ΣΥΠΑ, και ήμασταν εκεί πρόσφατα, όταν εξετάζαμε τα θέματα ιδιοκτησία ε, και ελέγχου. Εγώ είμαι υπέρ τη ελεύθερη αγορά. δεν έχω πρόβλημα ποιος είναι τη κάποιες εταιρείας κλπ. Έχουμε διάφορες προσεγγίσει για αυτά τα θέματα. Το ότι φτάσαμε τη ΣΥΠΑ στο 24% με κάνει να θαυμάζω. Ερώτηση. Πόσο χρόνο αφιερώνεται στι συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, όταν αναφέρθηκαν στι άλλε αγορέ αναδυόμενε. Θέλω να ξέρω περισσότερα γι' αυτά. Αναφερθήκατε στον Καναδά. Άλλη μεγάλη αγορά ο Καναδά. Σωστά αυτά που αναφέρατε. Μιλάμε για, μπορεί να μιλάμε σαν για ανταγωνισμό και συμφωνίες για υπηρεσίες κλπ. Αλλά αν δούμε ποια είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, υπάρχουν υψηλοί φόροι. Υπάρχει μεγάλο άχθος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ειδικό τέλος και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επιτρέπουμε σε χώρες να αποφασίζουν πώς θα αντιμετωπίσουν ε, το φόρο και ήταν και αποτυχία για τις σχέσεις ε, ε, το εμπόριο ρήπων. Και δεν ευνόησε το περιβάλλον. Άρα ελπίζουμε ότι η ΚΑΟ ίσως να βρει κάποια λύση. ο ουρανός, τον υποστηρίζω ένθερμα. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά το πώς κινούνται κάποια κράτη-μέλη. πως μενα αφουσιαμένα άλλα κράτη-μέλη, όχι το δικό μου. Έχουμε και το ΣΕΖΑΡ, την τεχνολογία, όλα όσα συνεπιφέρει ο νέος ουρανός. Θα περίμενα να κινηθούμε εκεί. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία λύση. Αν κάποιος στον πλανήτη πιστεύει αυτό το ισχύει, θα αποτύχουν. Ποτέ δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες, προσεγγίσεις, πλαίσια. Θέλουμε κάποια πρότυπα. Περιμένουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί όμως να επιβάλλει πάντα πράγματα σε τέτοιες χώρες. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε την αγορά. Εν γέννη, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, Πρόεδρε, να διεξαχθεί συζήτηση Πολλά ερωτήματα εκκρεμούν. Λείπουν πληροφορίες. Καλή τύχη στις συζητήσεις όσον αφορά τις συμφωνίες αυτές. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ανέφερα και τις άλλες χώρες. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτές. Ίσως πρέπει να ανέβουν σε προτεραιότητα. Κάθε φορά εδώ κουβεντιάζουμε το περισσότερο χρόνο της ΕΠΑ. Θέλουμε όμως και για άλλες χώρες περισσότερες πληροφορίες και πρέπει να καταβληθεί η δέουσα προσπάθεια. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Θα ήθελα να αναφερθώ, Πρόεδρε, σε κάτι που εισήγαγε και στην παρέμβασή του ο Σαΐντ Ελκαντράουι. Δηλαδή, όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι διάφορες εταιρείες. Ερώτηση. Το πλαίσιο των συμφωνιών, όπως παρουσιάστηκε, με πολύ θετικό τρόπο, επηρεάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές εταιρείες συγκρίση με τις εταιρείες των, α, της Ανατολής που επενδύουν, ανοίγουν νέες αγορές, νέα δρομολόγια κλπ. Και αποκτούν νέες μεταφορικές ροές. Α, πώς συγκρίνονται αυτές με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Γιατί υποφέρουν λόγω πολλών κανονιστικών περιορισμών και των συνθήκων της αγοράς. Όταν γίνονται οι προπολογισμοί ε, μάλλον όταν γίνεται ο απολογισμό βλέπουμε ότι χάνουν. Εάν δεν αλλάξει η προσέγγιση θα αυξηθούν οι απώλειες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ακριβέστερες, συστημικές ενδείξεις μέτρα που θα μπορούσε να θετήσει αυτό το κοινοβούλιο. Προσέγγιση. Θέλουμε να εξετάσουμε τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, με το Ισραήλ, με τις Αφρικανικές χώρες και άλλες, μεμονωμένα. Αλλά ίσως έτσι χάνουμε τη σφαιρική προσέγγιση, τη σφαιρική εικόνα μπορούμε να έχουμε στα βασικά σημεία αναφορά δύο-τρία που να μπορούμε να τα έχουμε υπόψη μα όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθούμε για τι διαπραγματεύσει. Μπένιον. Ωραία. Οπότε έμεινα εγώ τελευταίος. Θα ήθελα να τονίσω και εγώ αυτό που είπαν κάποιοι προλαλήσαντες Γιατί είναι το ότι συγκεντρωνόμαστε στη συμφωνία με τη, με τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά, τη Βραζιλία, σημαντικά είναι όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται με τη Ρωσία, με την Κίνα, Ινδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Τέσσερι γραμμέ αναφέρονται στην έκθεση. Με τη Σιγκαπούρη, τι γίνεται με όλε αυτέ τι χώρε και τι ε, αντίστοιχε συμφωνίε, προ τα που κατευθύνονται. Αναφέρθηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τι γίνεται εκεί γιατί βλέπω το περιφερειακό αεροδρόμιο του Μάντσεστερ που γνωρίζουμε κάλλιστα με την κυρία Φώστερ και το λατρεύουμε μέχρι θανάτου. Φαίνεται κάτι γίνεται στο, στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Βλέπουμε τις α, ε, ε, πτήσεις που κάνει Virgin α, ε, προς τη Φλόρινα, διατλαντικές, αλλά πού είναι η ITR, πού είναι το Κατάρ, πού είναι τα Εμμυράτα, η Σιγκαπούρη, η Air Continental. Βλέπετε τι εννοώ. Είναι όλες ε, ξένες, ε, μη κοινοτικές εταιρείες. Μόνο η Virgin έχει ε, μία πτήση από το περιφερειακό του Μάντσεστερ. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες στο Μάντσεστερ είναι ξεκινοτικές όπως είπε ο κύριος Καν, υπήρχε μια ιδεολειψία, μια έμονη ιδέα με το θέμα αυτό. Και αν ρωτήσει κανείς τους επιβάτες, οι περισσότεροι είναι ενθουσιασμένοι. Πηγαίνω στο Παρίσι, στο Σαλντεγκόλ και ακούω πολλά παράπονα για το Σαλντεγκόλ. Προσπαθώ να αποφύγω το Heathrow, προσπαθώ να μην περνάω καθόλου από εκεί. Και για τη Φραγκφούρτη ακούμε διάφορα. Οπότε με ενδιαφέρει η ιδέα σας. Επίσης, η υποβάθμιση των υπηρεσιών που είχαμε με τις διάφορες α, συμμαχίες. Και τι γίνεται με τις συνεργασίες αυτές. δεν ξέρω όταν θα φτάσει ο καιρό που δεν θα κλείνω καν στην με την Lufthansa, αλλά θα κλείνουμε κατευθείαν με τη Star Alliance. Αλλά όταν σας μίλησα για το Μάντσεστερ και την απελευθέρωση που γίνεται με, την, με τη ΣΥΠΑ, ναι μεν άνοιξαν δρόμοι, αλλά σίγουρα υποβαθμίστηκαν τα αεροσκάφη. Γιατί στο παρελθόν ε, πετάμε με 757 ε, σε διατλαντικές πτήσεις και δεν είναι και πολύ άνετες όταν χρειάζεται κανείς να, κάνει, να πάρει οικόνομη εισιτήρια και να πετάει με το προλαταριάτο, ενώ παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη άνεση οπότε υπάρχει και μια αρνητική πτυχή σε αυτή την απελευθέρωση και θυμάμαι και εγώ, θα θυμάστε και εσείς θυμάστε τον κύριο Καγιάκα τι καταπληκτική συμφωνία μας έλεγε ότι συνήψαμε με την ΙΠΑ. Α, κάλυψε ακόμη και τα όπλα. Καταπληκτική συμφωνία. Και κάποιος είπε ότι ε, γίνεται μια υποχώρηση προς τους Αμερικανούς ε, ευελπιστώντας ότι θα κάνουν αντίστοιχε υποχωρήσεις στο μέλλον και οι Αμερικανοί προς εμάς. Τελικά βλέπουμε ότι ο απολογισμός είναι αρνητικός. Δώσαμε εμείς λίγη μαρμελάδα, περιμέναμε από αυτούς, τελικά εμείς ε, βλέπουμε ότι δώσαμε πολύ περισσότερα από ό,τι πήραμε. Και τελικά αυτά που περιμέναμε δεν υλοποιήθηκαν. Πού πήγε ο κύριος Καγιάκ. Εξαφανίστηκε, έγινε καπνός και δεν ήρθε να μας πει γιατί δεν έγιναν αυτά που περιμέναμε. Βέβαια, μας είπαν κάποιοι ότι άλλες δυνατότητες δεν είχαμε στις διαπραγματεύσεις. Τότε μη μας λέτε, μη μας παραμυθιάζετε με το πόσο καταπληκτική ήταν η συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία, αλλά όχι ότι ήταν και τόσο καταπληκτική. Επίσης, το ενδιαφέρον με την έκθεση είναι ότι ουσιαστικά αποκαλύπτονται οι οι πόνοιές μας αρνητικές για τη συμφωνία με τις, για τις αεροπορικές μεταφορές. Δεν ξέρω. Αν έχουμε ένα σύστημα με επιδόσεις από το α είναι το καλύτερο και το ε είναι το χειρότερο, δεν ξέρω τι βαθμό θα βάζαμε. Πάντως, στην καλύτερη περίπτωση βάζουμε C ένα πολύ μέτριο βαθμό. Μπορεί να μην είναι ακόμη, να μην κόβεστε, αλλά σίγουρα οι επιδόση είναι πολύ μέτριες, οι βαθμοί είναι πολύ μέτρια. Κύριε Μπόλντεν, διαβάζοντας την έκθεση, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει μια ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση και αναθεώρηση. Ευχαριστώ, με προετοιμάσατε πολύ σωστά ε, είναι πολύ καλό που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά το σημαντικό αυτό θέμα. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την άριστη ε, έκθεση του κ. Μαρινέσκου. Αρκετά ενδιαφέροντα σχόλια ακούστηκαν και βλέπουμε πώς ενδιαφέρεται η Επιτροπή για το θέμα. Συνεχώς το συζητάμε. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα το πρωί είναι ενδιαφέρουσα. Παρουσιάστηκε άριστα και ευχαριστώ πολύ τεράστιος αριθμός θεμάτων που αναφέρθηκε. Και τα μέλη αναφέρθηκαν στον Ευρωπαϊκό Ουρανό και την ανταλλαγή λοιπόν το ETS, αλλά φαντάζομαι ότι ε, δεν έχω αρκετό χρόνο για να τα αναφέρω όλα αυτά. Θα περιοριστώ στην έκθεση λοιπόν. Διάλογος εδώ στο μικροφόνο. Γενικό σχόλιο. Θεωρούμε ότι η έκθεση είναι έχει πολύ αρνητικό τόνο. Και όσον αφορά τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όσον αφορά τι προοπτικέ. Και είναι άκρως αντίθετη σε σχέση με την ανακοίνωσή μας, που είναι στρατηγική ανακατάταξη και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίνουν τη θέση μας και την έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου, παρόλο που ακόμα τελεί υποσύνταξη το κείμενο. Στη σελίδα 72 λέει ότι η χρυσή εποχή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Αεροπλοίας έληξε. Και αυτή η εποχή χρονολογεί τη δεκαετία του 90. Παράξενο, διότι το 2003 μόλι αποφάσισε το δικαστήριο και προσθέτει και μια μυστηριώδη γραμμή ότι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν διευκολύνει θετικέ εξελίξει. Αυτέ λαμβάνουν υπόψη παρά την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Γιατί αναφέρονται αυτέ οι απόψει, εδράζονται επί κάποιων παραδόξων βάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την φήμη που έχουν οι συντάκτες του κειμένου. Λέει τα στοιχεία για συμφωνίες με γείτονες μοιάζουν ε, με τη κυκλοφορία με χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνία. Και ο κ. Πόψη είπε ότι κανένα από τα στοιχεία που έχουμε δεν δείχνει ότι έχουν σημαντική, σημαντικό αντίκτυπο οι ε, συμφωνίε. Αυτό είναι σημαντική κατηγορία αν λυθεύει. Παράδειγμα το Μαρόκο. Παράδειγμα. Κύριε παραθέσατε σαν παράδειγμα το Μαρόκο ότι δεν υπήρχε καμία επιρροή. Πριν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο η κυκλοφορία μεταξύ Ευρώπης και την Ισία ήταν δύο φορές από αυτή με το Μαρόκο. Όταν ετέθησε ισχύ η συμφωνία, έκτοτε, τώρα οι επαφές, οι συγκοινωνίες από 6,6 εκατομμύρια επιβάτες 2006 πήγε στα 11 εκατομμύρια 2011 όσον αφορά κυκλοφορία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Μαρόκου. Ενώ η συγκοινωνία, οι επιβάτε που μεταφέρονται μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία παρέμεινε σταθερό. Όφέλο οικονομικό είναι περίπου 3,5 δις. Μειώθηκαν οι ναύλοι μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου κατά 40%. Αυτά τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Άρα προβληματίζομαι, πραγματικά προβληματίζομαι όσον αφορά αυτά που αναφέρονται εδώ. Και κάτι άλλο που αναφέρθηκε. Ενδιαφέρονται. ΠΟΕ. Ήμου, είχα συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα. Βασική αρχή του ΠΟΕ είναι η αρχή της πλέον ευνοούμενης χώρας. Ό,τι προσφέρει σε έναν εταίρο προσφέρει σε άλλους εταίρους. Αυτή είναι η αρχή. Ο κ. Καν μπορεί να μας πει ότι αυτή την αρχή εφαρμόζει η ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις. Δεν νομίζω. Μέχρι τότε ο ΠΟΕ είναι ελκυστικό τόπο για διαπραγματεύσει όσον αφορά τι ε, υπηρεσίες αερομεταφορών. Γενική εικόνα. Άποψη που συμπίπτει με αυτή του Συμβουλίου. Και γι' αυτό μα δίνει νέε εντολέ Μα ζητά να δώσουμε νέε εντολέ για να προχωρήσουμε προ το χρυσού αιώνα, η χρυσή εποχή. Άποψη του Συμβουλίου ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Συμφωνώ με τον κύριο Καν. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια λύση για όλου. Στι διαπραγματεύσει βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν οι συμφωνίες που είναι ίδιες για όλου. Κάθε συμφωνία είναι διαφορετική και διακριτή. Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω, είπα. Επ' αυτού συγκεντρωνόμαστε. Πάντα θέλουμε περισσότερε διαπραγματεύσει. Αυτή η συμφωνία είναι ζωντανή. Πρόσβαση στην αγορά, ιδιοκτησία, Έλεγχο. Ευχαριστούμε που υποστηρίξατε σαν Επιτροπή στα θέματα ιδιοκτησία άλλα ρυθμιστικά θέματα συνεχώ είναι αντικείμενα διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ και μέσω τη μεικτή επιτροπή που ανέφεραν κάποιοι. Δοθέντω ότι εφαρμόσαμε τη συμφωνία και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω Καναδά εν το μέσο μια φοβερή ύφεση και οικονομική κρίση που ανέφερε και ο Σκαντράουι, Αλκαντράουι, είναι πολύ πρόημο τώρα να θεωρήσουμε ότι δεν θα έχουν αποτελέσματα τη συμφωνία. σω έχουμε και άλλη ευκαιρία όταν έχουμε τι διαπραγματεύσει FTA όπω ανέφερε η κυρία Μάισνερ και πριν βαθμολογήσουμε, ενδιάμεση βαθμολόγηση να δώσουμε στην, ε, ε, σε αυτό που ετοιμάζουμε. Η δίκαιο, ο δίκαιος ανταγωνισμός αναφέρθηκε από τον κύριο Καν, σημαντικότατο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα προωθήσαμε την αρχή αυτή. Στη διάσκεψη αερομεταφορές στο Μοντρεάλ, με μια νέα θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξανά θα το τονίσουμε στην επικείμενη συζήτηση με τις χώρες του κόλπου. Κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά κάποιες άλλες χώρες. Έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ζήτησαν προσέγγιση προσαρμοσμένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντί Τουρκία, Ινδία, Ρωσία, κάποιε χώρε του κόλπου, ΑΖΕΑΝ και όσο πιο γρήγορα γίνεται Κίνα. Το Συμβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει προσεγγίσει. Όχι για εντολή σε κάθε περίπτωση για διαπραγματεύσει, αλλά σε περισσότερε περιπτώσει. Θα σταματήσω. Μπορούσα να πω πολλά. Αλλά κλείνω με δύο δικαστικά αν επιτρέπετε. με τα μάλα. Διότι η DG Move είχε τη δυνατότητα να αντιθεί με τον κύριο Πρόπστ σε πρώιμο στάδιο των προσπαθειών. Θα χαιρόμασταν πολύ να συνεχίσουμε επαφέ μαζί, για, μαζί του για κάποια στοιχεία. Λυπούμεθα που δεν είχαμε την ευκαιρία. Από τον πρόλογο της εκθέσεως ακούγεται σοβαρή κατηγορία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει στο ε, Κοινοβούλιο ε, στα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων των μεικτών επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί για αυτές τις συμφωνίες. Ο κ. Πρόπιστη είχε πλήρη πρόσβαση στις εκθέσεις της Μικτής Επιτροπής. Θα ήταν καλό να αναφέρετε Εάν μας ζητούσε το Κοινοβούλιο επίσημα θα έπρεπε να ελέγξουμε σύμφωνα με τους κανόνες διαφανείας των γράφων, τι λένε τα κράτη-μέλη και τα συμβαλόμενα μέρη. Δεν είμαστε αποκλειστικοί διοικητές των εκθέσεων. Δεν είναι πρόβλημα για μας. Αν το Κοινοβούλιο θέλει να δει εκθέσεις της Μικτής Επιτροπής, πείτε το μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα δέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπόλτουιν. Ήθελα να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπα αφήστε την Επιτροπή να μιλήσει γιατί ήταν κάπως αρνητική η προσέγγιση της ε, εκθέσεων αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, μιλήσαμε ότι αυτό είναι κουταβάκι που δημιουργείται η προσπάθεια και συζητήσεις. Αν μεγαλώσει το κουταβάκι και γίνει σκύλαρος θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εκθέσεις αφορούσαν την έκθεση, εκθέσεις αφορούν τα μέλη. Κύριε Βάντενστάιν, αν θέλετε να ξεκινήσετε να προσπαθήσετε να δώσετε απαντήσεις σε κάποια θέματα που αφορούν εσάς και μετά ο κ. Πρόπ και ο κ. Καν θα συνεχίσει. Ευχαριστώ Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα δύο ερωτήματα που ετέθησαν. Συγκεκριμένα τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και τις ε, συμφωνίες. Το ζήτημα των επενδύσεων, παραδείγματος χάρη πρέπει να το δούμε ως ένα ζήτημα αριθμιστικής σύγκλησης. Προσπάθησα να το αναφέρω στις γενικές μου παρατηρήσεις και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρέπει να έχουμε μια καλύτερη κοινωνική συμφωνία μεταξύ των υπαλλήλων, ε, των πιλότων δηλαδή και στις δύο όχθες του Ατλαντικού και είναι κάπως παράδοξο δεδομένου του ότι οι πιλότοι αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί στην επικοινωνία και επαγγελματίες Νομίζω πως υπάρχει μια παράλληλη κατάσταση μεταξύ των πιλότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ. Δεν έχω μια μαγική λύση. Αλλά εάν οι πιλότοι βλέπουν κάτι θετικό στη δημιουργία συμβουλίων εργαζομένων στο επίπεδο συμμαχιών αεροπορικών εταιριών, θα έχουμε να έχουμε προσωστή κατεύθυνση, γιατί πρέπει και αυτοί να εμπλακούν. Και αν εμπλακούν, νομίζω πως οι ε, δυσκολίε θα είναι πολύ λιγότερε στη ΣΥΠΑ για τις επενδύσει Και εδώ πέρα έχουμε και το ζήτημα που ανέφεραν πολλοί ομιλητέ, το θέμα δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ, ε, μεταξύ αεροπορίας και λοιπόν κλάδων. Νομίζω πως οι νέες αυτές εμπορικές διαπραγματεύσεις πραγματικά παίρνουν μορφή. Καλό θα ήταν η απελευθέρωση των επενδύσεων να αντιμετωπιστεί με γενικό τρόπο για να συμπεριληφθούν πράγματα όπως οι αεροπορικές μεταφορές γιατί έτσι μπορούμε να εξορροπήσουμε και την απελευθέρωση του εμπορίου από άλλους κλάδους μη αεροπορικούς και έτσι θα μπορούσαμε να δούμε και κίνητρα στη ΣΥΠΑ για να αρθούν αυτά τα εμπόδια. Και το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε άλλες σχέσεις, αναφέρθηκε το ζήτημα των προβλημάτων με χώρες ε, όπως η ανάγκη να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποτελεσματικά σε προβληματικές καταστάσεις, όχι οπωσδήποτε να πάμε σε μια πλήρη συμφωνία, απλά για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Και αν μπορούμε νομίζω να αντισταθμίσουμε και άλλα εμπορικά ζητήματα, για να υπάρχει κάπου αλλού αντισταθμίζαμε, νομίζω μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Δηλαδή το να περιοριστούμε στην αεροπορία δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μουχλούς πίεσης. για να επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θετικά ή αρνητικά. Νομίζω πως... Βασικά αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέθηκε ερώτηση για Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ε, Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτείων. Όπως σας είπα το διμερές πλαίσιο δεν επιτρέπει να πείσουμε μια χώρα που δεν θέλει να κάνει υποχωρήσει να τις κάνει. Όντως, κυρία Φώστερ, υπάρχουν συμφωνίες και χώρες με κάποιες συμφωνίες, όχι πολλές. Τι γίνεται όμως με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Κορία. Δεν θέλουν οι χώρες αυτές σε διαπραγμάτευση. Μπορεί να πει ότι θέλει το Συμβούλιο και να δώσει εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί, αλλά οι χώρε αυτέ είναι απρόθυμε για διαπραγμάτευση. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη ΣΥΠΑ μπορεί να είναι καλό φόρουμ για να πούμε θέλουμε να μιλήσουμε και για την αεροπορία. Και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε αυτό και αυτό. Αν πούν όχι, τότε θα αφαιρέσουμε κάτι από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, κάτι που επιθυμούν εκείνε. Γίνεται ένα, μια δοσοληψία στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορία έχουμε τον κανόνα Most Favored Nation. Αλλά αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2002, δεν έχουμε άλλη λύση. Ή τουλάχιστον κάποιες διμερείς συμφωνίες με ορισμένες χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι στις διμερείς συμφωνίες δεν έχουμε αρκετούς μηχανισμούς. Ένα σημαντικό μηχανισμό Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου είναι το σύστημα διαιτησία. Όταν μια χώρα λέει θα δεσμευτώ γι' αυτό και μετά αθετεί τις υποχρεώσεις, τότε συγκροτείται ένα πάνελ και η απόφαση του πάνελ είναι υποχρεωτική για τη χώρα αυτή. Όταν πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο φόρουμ, ε, θα έχει συνέπειες για, την, για τον ευρωπαϊκό κλάδο. Και αν ο κλάδος δεν ε, είναι ικανό να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, τότε θα το πρέπει να το αποφύγουμε και να, να θέσουμε άλλους στόχους, φιλελεύθερους ή προστατευτικούς αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε με, τη, τον κλάδο. Αν πει ο κλάδο θέλουμε άνοιγμα, είναι σε θέση να το υποστεί όμω αυτό το άνοιγμα. Επίση, ό,τι αφορά την κανονιστική σύγκληση, κατά τη γνώμη μου, το ότι βάλαμε στι διμερεί συμφωνίε κάποιε διατάξει για τα δικαιώματα κυκλοφορία ήταν λάθο. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να μιλήσουμε για κανονιστική σύγκληση με του εταίρου, πέραν των δικαιωμάτων αυτών έχουμε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά, τη Βραζιλία, τη Ρωσία και με την Κίνα για, τον για την κανονιστική συγκλήση ότι αφορά την ε, εναέρια ασφάλεια. Κάποιες χώρες έχουν αεροναυπηγική και θέλουν ε, έχουν συμφέρον να έχουν πιστοποίηση τα σκάφη τους για να πολιούνται παντού. Οπότε αντί να δημιουργηθούν προβλήματα στην πιστοποίηση των αεροσκαφών, θέλουμε κανονισμούς που θα είναι σχετικά και διατάξεις που θα είναι σχετικά ε, συγκλίνουσες, ώστε όταν λαμβάνει κανείς πιστοποιητικό σε μια χώρα να μπορεί εύκολα να πουλήσει το εμπόρευμά του και το αεροσκάφος του και αλλού. Και το γεγονός ότι ε, συνδέσαμε την κανονιστική σύγκληση με τα δικαιώματα κυκλοφορίας ε, δημιουργεί πρόβλημα και τη μία περίπτωση και στην άλλη, και στην κανονιστική σύγκληση και στα δικαιώματα αυτά. Μερικοί λένε ότι από τις ε, συμφωνίες κάποιοι βγήκαν κερδισμένοι, γιατί κάποιες χώρες δεν είχαν κάνει συμφωνία, είχαν λίγα δικαιώματα. Όντως υπάρχουν κάποια δυνητικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις συμφωνίες. Είναι χρήσιμα όμως αυτά. Γιατί μια χώρα δεν είχε συνάψει συμφωνία με τη ΣΥΠΑ γιατί δεν είχε συμφέρον, δεν είχε αεροπορικές συνδέσεις ούτε είναι σίγουρο ότι κέρδισε κάτι. Υπάρχει ένα δυνητικό πλεονέκτημα. Το θέμα είναι αξιοποιηθεί και αυτό το πλεονέκτημα. Εγώ από τα στοιχεία που έχω διαπιστώνω ότι δεν αξιοποιήθηκαν τα πλεονεκτήματα αυτά. Ο κύριος Μπάλτον λέει, α, κοιτάξτε ότι στο, στο Μαρόκο είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά απάντησα ότι ναι, αλλά από το 2001 είχαμε καλή ε, καλέ εξελίξει, Γιατί από το 2001 τροποποίησε άρτην το Μαρόκο την ε, πολιτική ε, στην αεροπορία. Μέχρι τότε είχε προστατευτική πολιτική, προστάτευε την Air Royal Μαρόκο. Μετά σκέφτηκε ότι ο τουρισμό είναι πιο σημαντικό. Οπότε μόνο μέρο έκανε ένα άνοιγμα προ όλε τι κατευθύνσει. Όλε οι αεροπορικέ εταιρείε που θέλουν να διασυνδέσει με το Μαρόκο έχουν δικαίωμα να τι εφαρμόσουν. Γι' αυτό βελτιώθηκε η κατάσταση στο Μαρόκο. Αν είχε κρατήσει την παραδοσιακού του πολιτική του Μαρόκου, δεν θα είχε διαπραγματεύσει και διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε τέτοια συμφωνία γιατί τροποποίησε άρδιν την πολιτική του το Μαρόκο. Οπότε, τι γίνεται, αν θέλουμε συμφωνία με την Κίνα, τι θα γίνει, τι θα λάβουμε ως αντιστάθμισμα ή με τους Ρώσους. Είπαμε στους Ρώσους κάποια στιγμή, σταματήστε να ζητάτε ρόγελ τη για την υπέρπτυση από τη Σιβηρία. Είναι πολλά τα χρήματα που πηγαίνουν στην Αεροφλότ και ίσως και αλλού. Και τους λέμε, ότι αυτή την περίπτωση δεν θα γίνεται μέλος του ΠΟΕ. Ε, έκαναν μια προσπάθεια, είναι μέλη του ΠΟΕ, αλλά ακόμη συμφωνία δεν είδαμε. Αν τέτοιες συμφωνίες ε, τις κάνουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ, μπορούμε να ζητήσουμε ένα πάνελ του ΠΟΕ για να καλέσουμε τον εταίρο να τηρήσει μια δέσμευση. Είπατε ότι δεν έχετε πρόσβαση στα πρακτικά των ε, μεικτών επιτροπών. Τα ζήτησα και μετά από τρεις μήνες μου απάντησαν «Ελάτε, θα σας καλέσουμε στη συνεδρίαση, θα σας τα δείξουμε, παρουσία μας μπορείτε να τα κοιτάξετε, αλλά δεν μπορούμε να σας τα στείλουμε». Μπορείτε να ξανάρθετε αν θέλετε ή να μας στείλετε ερωτήσεις. Χρειάστηκα τρεις μήνες για να μπορέσω σε ένα γραφείο να διαβάσω μερικά από τα πρακτικά των μεικτών επιτροπών. Αυτό δεν είναι πρόσβαση ελεύθερη. Και προσπαθώ να δω αν οι συμφωνίες που έχουν ε, συνεχθεί είχαν κάποια θετικά αποτελέσματα. Και βλέπετε σε τι συμπεράσματα κατέληξε. Δεν βλέπω και μεγάλη διαφορά. Και από μερικά πρακτικά μεικτών επιτροπών διαπίστωσα ότι δεν ε, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις ε, για την κανονιστική σύγκληση και πολύ λυπούμε. Πολύ ευχαρίστω να ξαναδώ τα πρακτικά, αλλά δεν νομίζω ότι μου διέφυγε τίποτα τη προσοχή μου από μια πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ κύριο Χάν. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρκετές ε, ερωτήσεις αφορούσαν εμένα. Θα τις διατρέξω μία-μία και ελπίζω να μην λησμονήσω κάποια. Αν το κάνω θυμίστε το μου. Για την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ε, στον ΠΟΕ. Μαζί με το ερώτημα που έθεσε ο κ. Μπόλτουιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποια θα ήταν θέση του ΠΟΕ για να συμπεριληφθεί σε αρμοδιότητε του και στην εντολή το θέμα των αερομεταφορών, το μέσο των αερομεταφορών αποκλείεται ρητά από τη διαπραγματευτική, ε, από την εμπορική εντολή του ΠΟΕ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τεθεί, να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις και τομέας σε επίπεδο ΠΟΕ, αλλά μας, ε, μας αρέσει καλύτερη η λύση αυτή η μεικτή επιτροπή και συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως ΕΙΠΑ όσον αφορά τις ε, αερομεταφορές υπηρεσίες. Αν πάμε στον ΠΟΕ, μπορεί να γίνει αυτό μακροπρόθεσμα μετά από δεκαετίες. Ο ΠΟΕ μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να έχει πλήρεις αρμοδιότητες και τις αερομεταφορές για την ώρα όμως σαν τομέας είμαστε ικανοποιημένοι με τον ΙΚΑΟ να καλύπτει το θέμα. Και κάτι που θα θέλαμε θα ήταν να αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ασφάλεια και τεχνική συνεργασία να έχουμε αρμοδιότητα για θέματα ιδιοκτησίας και ελέγχου. Για την ερώτηση του κυρίου Ελχαντραουή για την γρήγορη ολοκλήρωση των ε, διαπραγματεύσεων. Πράγματι, έχει κάποια αξία αυτό. Για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη το ε, εάν είναι θετική ή αρνητική, αλλά να είναι ρεαλιστική για το τι θέλουμε τώρα να έχουμε με τις ε, συμφωνίες αυτές. Και το πρόβλημά μου είναι πως ε, τείνουμε να τα παρουσιάζουμε τα πράγματα θετικά αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, ποιες είναι οι συνθήκες για την ιδιοκτησία, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ελευθερία και έτσι, να δούμε αν ε, θα έχουμε καλύτερη κατάσταση για, την τον ευρωπαϊκό κλάδο. Και δεν είναι αυτό πάντα σε πρώτο πλάνο. Και αν συμπεράνουμε πως είναι θετικά τα πράγματα, τότε είναι καλό αυτό, ναι. Για τις συμμαχίες και για το εάν ε, μπορούν να σημαίνουν κάτι. Εντός των ε, συμμαχιών, ε, κοιτάξτε, αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που έχουν ε, εξαίρεση από τους κανόνες του ανταγωνισμού και στις δύο όχθες του Ατλαντικού ε, για την βέλτιστη χρήση της αγοράς. Δεν βλέπω πώς θα μπορούσαν έτσι γρήγορα να αξιοποιηθούν στο πολιτικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ εμπορικές ε, στον προσανατολισμό τους. Είναι κάποιες ενώσεις όπως η αντίστοιχη της δικής μας ε, στην Ουάσιγκτον, η A4A, που κοιτάνε να δουν το τι γίνεται με τις ε, συμμαχίες. Κύριε Μάισνερ, νέοι ναι, τύποι συμφωνίων. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που θα δούμε στο μέλλον είναι πολύ περισσότερες συμφωνίες κατά περίπτωση. Τα θέματα που θα συζητούμε θα μοιάζουν πολλά με αυτά που συζητάμε σήμερα σαν Ευρώπη με μη ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ίσως πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί και πιο δημιουργικοί όσον αφορά τα δικαιώματα κυκλοφορίας που θα θέλαμε να διαπραγματευτούμε. Θα έπρεπε ίσως να συμπεριλάβουμε αυτό που είπαν κάποιοι θέματα εργασιακά και μη εργασιακά. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε περιβαλλοντικά θέματα στις συμφωνίες. Υπάρχουν αρκετές συμφωνίες που έχουμε συνάψει που αφορούν το θέμα ασφαλείας των επιβατών, ασφαλούς λειτουργία των αεροσκαφών, τα δικαιώματα των επιβατών κλπ. που συμπεριλαμβάνονται. Θα πρέπει να ετοιμάζουμε συμφωνίε κατά περίπτωση πιστεύω και όχι μια ενιαία προσέγγιση. Αυτό που είπε η κυρία Φώστερ. Πέρα από Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία κλπ. Έχουμε Μολδαβία, Αζερβαϊτζάν, ε, ε, πληθώρα κρατών με διάφορες ιδιαιτερότητες, ε, κάποια χαρακτηριστικά, κάποια μας ικανοποιούν, κάποια όχι. Άρα χρειάζεται να γίνεται πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση πριν διαμορφώσουμε μια σφαιρική πολιτική. Και τέλος, αυτό που αναφέρατε, Πρόεδρε, λυπούμε, διότι δεν υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι αερομεταφορές, σαν IA δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. να το θέσετε με τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες θα έλεγα. Αυτές είναι εμπορικές αποφάσεις και εγώ δεν μπορώ έτσι ανοιχτά να αναφερθώ εκτενώς σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Φώστα έχει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Θέλω να αναφέρω κάτι που αφορά τον κύριο Πρόπστ και τον συνάδελφό του. Εδώ αισθάνομαι ότι δεν θέλω πια να ζήσω ακούγοντα το που, βλέποντα που πάμε αυτέ τι συμφωνίε. Αρνητική ατμόσφαιρα, αρνητικότητα, φοβερά προβλήματα ακούω. Ρωτήσαμε τι γίνεται με Κίνα, Ρωσία και άλλου. Δεν θέλω λεπτομέρειε. Του μιλάτε. Αυτό θα μια απάντηση. Προφανώ αυτό θέλετε να πείτε. Μετά λέτε. Είναι θέμα των πιλότων αυτό με την Αμερική. Όχι, δεν έχει σχέση με του πιλότου και μόνο. Αν δεχόσαστε ότι όλα εξαρτάται από του πιλότου, Είναι τρέλα να σκέφτεται κανείς κάτι τέτοιο. Είναι το κογκρέσο, είναι τα διάφορα συμφέροντα που επηρεάζουν την κατάσταση. Τέλος. Σαν να γίνεται μάχη εξουσίας εδώ. Εσείς εκεί και η DG Move απ' την άλλη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι μάχες για την εξουσία. Χαίρομαι που δεν είμαι, δεν ελέγχω, δεν διοικώ κάποιο Ευρωπαίο αερομεταφορέα. Έχω ελάχιστη εμπιστοσύνη σε αυτά που κάνετε με αυτά που ακούω, για να είμαι ειλικρινής. Προτείνω λοιπόν να συμμαζευτείτε. Δεν με ενδιαφέρει αν συμφωνείτε, διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τη DG Move κλπ. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Πιάστε κουβέντα μεταξύ σας, βρείτε τα, βρείτε τα. Και όταν έρχεται, έρχεστε στην Επιτροπή για κάνα δύο σας επιτρέπουν, να μας δώσετε κάτι επικοδομητικό. Πλήρες, θετική προσέγγιση. Τι μπορείτε να κάνετε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν δυσκολίες, αυτό το καταλαβαίνουμε. Τι θα κάνετε όμως για αυτές. Αυτό είχα να πω και ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν διαδικαστικό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ο Πρόεδρος δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να αντιδράσει σε αυτά που υπόθηκαν. Όχι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό που είπε και ο Σβάντενστάινεν. Η δική μου εμπειρία με το Κογκρέσο ποια είναι. Ότι τρέμουν τα συνδικάτα. Αυτό είναι. Τώρα, φταίει το Κογκρέσο, δεν φταίει. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν μέρη υπερασπίζομαι αυτά που είπατε εσείς κύριε Βαντενστάινεν. Καλώς, ευχαριστώ και τους τρεις σας για την συνεισφορά σας στη συζήτηση. Ευχαριστώ που ήρθατε, που κάνετε τις παρουσιάσεις. Ευχαριστώ και τα μέλη. Στις 3 το απόγευμα θα τα πούμε για τη δράση για τον τουρισμό και το πρόγραμμα το σχετικό. Θα τα πούμε το απόγευμα λοιπόν. Καλή σας όρεξη.